Well, friends, we'll start uh, this meeting. Αγαπητοί φίλοι, ξεκινάμε αυτή την ε, δημόσια ακρόαση για τους ε, πρόσφυγες κοινωνική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ όλους. Κάποιοι από σας μάλιστα ταξιδέψατε μακρύ δρόμο για να είστε μέχρι τις Βρυξέλλες. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς ήρθατε και εσείς ε, Λίλιβοι που στα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Ε, αυτή είναι η κύρια, συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Σύστημα σε κάθε επίπεδο και προφανείς λόγους μας απασχολεί διότι μπορούμε να διαπιστώσουμε πως είναι όλους εξαιρετικές οι ανάγκες, όλους εξαιρετικές οι πιέσεις ε, που ασκούνται στους πρόσφυγες, όλους εξαιρετικές οι πιέσεις που ασκούνται στα κράτη-μέλη επίσης. Και την κρίση, την προσφυγική δεν την έχουμε αντιμετωπίσει με τρόπο ούτε ενιαίο, ούτε θα έλεγα καν ανθρώπινο μέχρι τώρα. Εξού και θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το σεμινάριο, τη δημοσιακή γιατί θα ακουστούν διαφορετικές φωνές. Θα ακουστούν οι φωνές των ειδικών. Θα ακουστούν οι φωνές που θα μας περιγράψουν την πραγματικότητα πως έχει αυτή τη στιγμή στην προσφυγική κρίση. Και βεβαίως θα μας πείτε και το τι συμβαίνει αφού έχουν φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρόσφυγες. Ευθύνη. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ένα καλό αποτέλεσμα. Καλές προτάσεις. Στην ακρόαση. Υπεύθυνοι πάντως να μας ε, κρατήσει στην ε, συζήτηση αυτή και να την ε, τοποθετήσει σε ένα πλαίσιο είναι ο κύριος Μπράντο Μπένιφάι από τους σοσιαλιστές και εισηγητής ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Μπένιφάι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εκλεκτούς μας διρογνώμονες οι οποίοι βρίσκονται εδώ στη συνεδρίασή μας αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας προκειμένου να μοιραστούν τη γνώση τους ε, μαζί μας. Όπως είπε και η Πρόεδρος, εγώ έχω διοριστεί εισηγητής ε, όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των μεταναστών, των προσφύγων και θα συντάξω μια έκθεση και μάλιστα έχω ολοκληρώνω αυτή τη στιγμή το πρώτο σχέδιο της έκθεσης αυτής στις 22 ε, Φεβρουαρίου θα ασταλεί το έγγραφο αυτό για μετάφραση και θα το παρουσιάσω εδώ στην Επιτροπή μας στις 16-17 Μαρτίου. Επίσης, υπάρχουν και επιτροπές οι οποίες ε, γνωμοδοτούν. Η Επιτροπή Πολιτισμού συγκεκριμένα πρόκειται να γνωμοδοτήσει για το ζήτημα της ε, πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής διάστασης. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ακριβώς ποια στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια θα εντάξω στην έκθεσή μου αυτή. Θα ήθελα και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των εκλεκτών καλεσμένων μας και είμαι σίγουρο ότι θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και ότι οι παρουσιάσεις αυτές θα μας εμπνεύσουν προκειμένου να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας. Σίγουρα το ζήτημα δεν είναι καθόλου εύκολο, αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι μόνο επειδή έχει μια έντονα πολιτική διάσταση, ή για να το θέσω λίγο πιο ουδέτερα, βρίσκεται στην ε, πρώτη γραμμή των ε, εθνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρόκειται παράλληλα και για ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευρύ, το οποίο καλύπτει την πολιτική ασύλου, τη διεθνή προστασία, ζητήματα αγοράς εργασίας, φορολογικά, δημοσιονομικά, μακροοικονομικά ζητήματα και θίγει επίση και το ζήτημα των διακρίσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν κάπω δύσκολο να καταφέρω να συντάξω ένα έγγραφο το οποίο θα μπορούσε να καλύψει με τρόπο γραμμικό όλα αυτά τα ζητήματα, καθότι έχουμε μια κατακαιρματισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τα ζητήματα αυτά και παράλληλα έχουμε μια περιορισμένη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς αυτούς. Πράγμα το οποίο κατέστησε την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού ιδιαίτερα ετερογενή. Από την άλλη έχω ένα συνδυασμό προγραμμάτων, συστημάτων, ταμείων, πολλά διαφορετικά τέτοια συστήματα, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο όλα αυτά τα πολυσχηδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με, με την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ σε κάποιες ε, βασικές εκτιμήσεις τις οποίες βασίζει η εκθεσή μου. Πρώτον, η προσφυγική κρίση είναι καταρχάς μια ανθρωπιστική κρίση. Κατεπηγόντως λοιπόν πρέπει να ανταποκριθούμε στην κρίση αυτή. Δεύτερον, το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι μία διαδικασία αρκετά δυναμική, αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία για μας και θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, τα κράτη-μέλη, αλλά και οι ε, οργανώσεις εκπροσώπησης των προσφύγων να συμβάλλουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να αναλάβουμε δράση πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς, προκειμένου να επιτύχουμε μια αποτελεσματική κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Τέταρτον, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, αυτό που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποια εναλλακτική λύση. Πρέπει ουσιαστικά να κινηθούμε σε αυτό το δρόμο. Αυτά είχα να σας πω εν είδη εισαγωγή και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπενιφέλη. Έχουμε έξι προσκεκλημένους εδώ που θα κάνουν τις δικές τους ε, τοποθετήσεις στη συζήτηση. Η κυρία Χάλα Ακάρη από τη Συρία. Εθνική Ένωση Προσφύγων και πρωτοβουλία των πολιτών του Μαρίεστατ της Σουηδίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε και σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα 8 με 9 λεπτά, θα ήταν τέλειο. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπενιφάη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με προσκάλεσε σε αυτή τη δημόσια κρόαση να μιλήσω για την ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμη η δική μου η παρέμβαση. Ως μέλος της Ένωσης Προσφύγων από τη Συρία και ως άνθρωπος που εργάζεται στην πόλη της ε, Μαρίενστατ της Σουηδίας για το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Θα ήθελα ιδιαίτερα σήμερα να αναφερθώ στα κύρια προσκόμματα ως προς τη διαδικασία της ενσωμάτωσης και να προτείνω κάποιες λύσεις και καλές στρατηγικές και δράσεις. Θα ε, αναφερθώ στο σουηδικό μοντέλο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα κράτος το οποίο αναλαμβάνει τις ευθύνες του εξ αρχής σε σχέση με τους πρόσφυγες και βλέπω πολλές ομοιότητες μεταξύ του σοηδικού μοντέλου και αντίστοιχα των πρακτικών που ακολουθούν άλλες χώρες, γι' αυτό ακολουθώ αυτό το πρότυπο, ε, το οποίο προσφέρει και την ε, άμεση κάλυψη σε στέγη ε, των των το άσυλο, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται η αίτηση ασύλου. Στην συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν να κοιτάξουν την πιο μόνιμη στέγη και ένα πρόγραμμα για ενσωμάτωση με τη δυνατότητα για εκμάθηση της γλώσσας και ανάληψη ε, επαγγελματικών δραστηριοτήτων εξεύρεστες εργασίες. Μπορεί να κρατήσει μέχρι και δύο χρόνια διαδικασία η οποία δεν ε, εκτελείστε πάντοτε απρόσκοπτα τόσο όσο μπορεί να φαίνεται. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν μακρές περίοδοι αναμονής μέχρι ότου εξεταστούν οι αιτήσει ασύλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτή την εποχή, μέχρι και δύο χρόνια μπορεί να περάσουν, ε, περίοδος κατά την οποία ο πρόσφυγας διαμένει σε καταβλισμούς με σοβαρό πρόβλημα υπερπληθισμού έξω από τις πόλεις. Πριν να πάρει λοιπόν την άδεια παραμονής, ο, η, πρόσφυγας δεν έχει δυνατότητα πρόσβαση ούτε σε μαθήματα γλώσσας, ούτε σε άλλη εκπαίδευση που μπορεί να προσφέρουν οι κρατικές δομές και βέβαια δεν εύκολη ζωή στους καταβλισμούς. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρόσφυγας. Ε, τον κάνουν να χάσει τον ενθουσιασμό του και την βούληση για μια νέα εκκίνηση. Και άρα περιορίζουν και τη δυνατότητα ε, αποτελεσματικής ολοκλήρωσης κοινωνικής ενσωμάτωσης στο μέλλον. Για τους πρόσφυγες που έχουν ε, υψηλότερη εκπαίδευση δεν υπάρχει δυνατότητα της επικύρωσης των ε, επαγγελματικών και πανεπιστημιακών πτυχίων και άρα δεν ε, δυσκολεύεται ιδιαίτερα η δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση. Η προσφορά θέση εργασία είναι πολύ περιορισμένη. Μόνο όσο υπάρχει επιδότηση από τι κοινωνικέ υπηρεσίε ε, κατά 60 με 70% και μάλιστα για το μέγιστο διάστημα ενό έτου ο εργοδότη είναι διατεθειμένο να προσλαμβάνει πρόσφυγε. Ε, Βεβαίω ο πρόσφυγα, ο εργοδότη πολλέ φορέ διστάζει και αποφεύγει να προσλάβει ε, ε, πρόσφυγες γιατί θεωρεί ότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει προβλήματα ή μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα επαφών ή πιέσεων και από ακροδεξιέ ομάδε. Έχουμε δει να διαπράττονται και εγκλήματα μίσου στου βάρου των προσφύγων. Φαντάζομαι θα αντιλαμβάνεστε πόσο επηρεάζουν αρνητικά όλα αυτά τη διαδικασία τη ενσωμάτωση. Οι πρόσφυγε έχουν ήδη το δικό του βαρύ φορτίο πόνου, έχουν χάσει τη χώρα του, έχουν χάσει του δικού του, έχουν περάσει μέσα από πάρα πολλού κινδύνου για να φτάσουν μέχρι τα σύνορα τη χώρα και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι κάνουν δηλώσει πω οι πρόσφυγε θα εξαναγκαστούν να επανέλθουν, να επανέλθουν στις χώρες τους μόλις επιληθεί η πολιτική κρίση και αντίστοιχα. Άρα λοιπόν έχει πάντα έτοιμη τη βαλίτσα του ο πρόσφυγας, ε, την κοινωνική ενσωμάτωση την αντιμετωπίζει μάλλον σαν περιττή πολυτέλεια. Και όταν ακόμα αποφασίσει να μπει μέσα στην κοινωνία, είναι τόσο διαφορετική σε κάθε τι αυτή η νέα κοινωνία και στο στάδιο αυτό ε, του γεννώνται φόβοι, ανησυχίες έχει ανάγκη να εκφράσει τις ανησυχίες αυτές, ε, να, να έχει κάποιον να τον ακούσει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό η ενσωμάτωση, η μετανάστευση ε, να συνεργαστούν αυτοί που είναι αρμόδιοι δηλαδή για τη χάραξη πολιτικής στα δύο αυτά πεδία, να φτιάξουν ένα σχέδιο μακρόπνο που θα καλύψει περίοδο πολύ μακράν του ασύλου και ε, τα μαθήματα της γλώσσας θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για την ε, διαδικασία της ενσωμάτωσης και βέβαια μεγάλη επένδυση. Η κοινωνία των πολιτών προσπαθεί να καλύψει από πλευρά τη ε, τα κενά, να συμπληρώσει το έργο των αρχών με μαθήματα γλώσσας, πολιτιστικές ε, δραστηριότητες, επικοινωνία με τον πρόσφυγα και τον ετούντα το άσυλο, γιατί προσεγγίζει και τον ετούντα το άσυλο. Θα είχα πάρα πολλά παραδείγματα να σας αναφέρω, αλλά δυστυχώς δεν θα μου φτάσει ο χρόνος μου από ό,τι βλέπω αλλά πρέπει να επισημάνω πως η κοινωνία της Νιστάτ και πολλών άλλων πόλεων κάνουν πολλά πράγματα για να ε, καλωσορίσουν αυτούς ε, τους ε, νεοφερμένους και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το, ότι υπάρχει αυτή η δουλειά είτε των ιδιωτών είτε των οργανώσεων για τους νεοφερμένους. Στα θέματα εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες απασχόλησης, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ανεργίας και ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω μελέτη ε, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα ανάπτυξη ενός σχεδίου για το χώρο εργασίας με υποστήριξη ε, για χαμηλότερη ε, αμοιβή έτσι ώστε να προσελκυθεί και ο εργοδότης ε, με ταυτόχρονη όμως υποστήριξη και σε επίπεδο γλώσσας και άλλων γενικότερων γνώσεων, έτσι ώστε μέσα σε δύο-τρία χρόνια ο εργαζόμενος πρόσφυγας να έχει αποκτήσει όλα αυτά τα εφόδια ώστε να μπορεί να εργαστεί σε υψηλότερο επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στην περίοδο που εκκρεμεί η αίτηση ασύλου για να κερδίσουμε χρόνο. Η αγορά εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνει ε, να, να αξιολογεί τα επαγγελματικά προσόντα ε, να μην επιβάλλει πολύ αυστηρά προγράμματα εκμάθηση εξ αρχής. Οι δημοτικές αρχές έχουν διάφορα προγράμματα, σχέδια για διαπολιτισμικό διάλογο, στα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν ε, και να διαλέγονται και οι πρόσφυγες μέσα από ένα συμβουλευτικό ίσως όργανο με εκπροσώπους τους, το οποίο θα, συνέ, συνέρχεται μαζί με πολιτικούς και εκπροσώπους των τοπικών αρχών ε, τακτικά έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές οι ανάγκες ε, ε και πολιτισμικές των νεοφερμένων. Οι νεοφερμένοι αυτοί και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι μικρότερα τα προβλήματα σε, σε μικρές πόλεις σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Πρέπει λοιπόν να γνωριστεί ότι είναι ύστερα από αυτό το τεράστιο κύμα ε, μεταναστών που έχουν φτάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι κατανοητό το ότι υπήρξαν κάποιε αντιδράσεις, οι οποίε είχαν καταγραφεί στη δεκαετία του 90 αντίστοιχα με την αφήξη των Βοσνίων στη, ε, στη Σουηδία. Μπορεί να δει κανεί τίτλου αντίστοιχου ε, στι εφημερίδε της εποχής μας με αυτές τις δεκαετίες του 90, αλλά ταυτόχρονα οι Βόσνοι είχαν αναγνωριστεί ως κάτι το θετικό για κάθε τομέα της, ε, του δημόσιου βίου στην Σουηδία ε, και τώρα πια είναι πλήρως ενσωματωμένη. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τις απαντήσεις στα ερωτηματικά. Μετά το διάλογο έρχεται η κατανόηση, η κατανόηση διαφορών όπως και ομοιοτήτων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι προκλήσεις ε, θα μας φέρουν όλους μαζί στην ίδια γραμμή για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα. Η Σύριοι σήμερα, η σήμερα και οργανώνονται και ε, συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών με κάθε δυνατόν τρόπο. Οι κοινωνίες οι τοπικές βοηθούν και ανταποκρίνονται. Συχνά έρχονται να μας ακούσουν οι πολίτες ε, όταν μιλούμε για μας, για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας. Βλέπουν ότι προσπαθούμε να ε, χτίσουμε και να αναπτύξουμε τη ζωή μας εδώ στην Ευρώπη, έστω και αν οι μας ήταν κάπου αλλού. Και θέλω να σημειώσω κλείνοντας κάτι πολύ σημαντικό. Ο πόλεμος στη Συρία δεν αμφισβητεί μόνο τις κρατικές δομές και την ύπαρξη των σύρων, αλλά κάθε έννοια αξιών. Εμείς στραφήκαμε προς την Ευρώπη λόγω του υψηλού επίπεδου των αξιών της και του σεβασμού προς τα δικαιώματα. Γι' αυτό αναμένουμε να διαδραματίσει η μεγαλύτερο ρόλο η Ευρώπη και στο Συριακό, αν όχι ε, σε θέματα συγκρούσεων τουλάχιστον ανθρωπιστικά. Η πόλη της Μαντάγια είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα υποφέρει ακόμη, η πολιορκία έχει φέρει το λοιμό, έχει φέρει το θάνατο και συνεχίζεται ακόμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μια τραγωδία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα χάρη στην υλοποίηση των αξιών, των αξιών για τις οποίες είναι η η Ευρώπη και οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και έξω από αυτήν. Σας ευχαριστώ. Thank you. <coughs> Εγώ σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Κάρη. Επόμενος ομιλητή, είναι ο δόκτωρ Wolfgang Miller, συντονιστής για τη μετανάστευση, task force για το άσυλο και ε, τους πρόσφυγες και από τη Γερμανία στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόληση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσει τη μητρική μου γλώσσα, λέει ο Μίλλερ. Ich vertrete eben die ο ΑΕΦ της Γερμανίας. Ε, ταυτόχρονα είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου όλων των ε, δημοσίων υπηρεσιών ε, εύρεσης εργασίας. Αλλά θα περιοριστώ στην κατάσταση που έχουμε στη Γερμανία. Για να δει κανείς τι γίνεται στην ένταξη στην αγορά εργασίας θα πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά εκείνων που πρέπει να ενταχθούν και να εσωματωθούν σε μια αγορά εργασίας. Θα σας αναφέρω σύντομα τα στοιχεία για τη Γερμανία. Έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους που χρειάζονται προστασία και που έφτασαν το 2015 στη χώρα. Αν θεωρήσουμε ότι χρειάζεται προστασία 50%, και κοιτάξουμε τι σημαίνει αυτό το ποσοστό εκείνων που είναι σε ηλικία ε, που να μπορούν να εργαστούν, παραγωγική, ε, είναι το 70%. Άρα θα πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 350.000 νέοι εργαζόμενοι. Εξ αυτών το 80% έχουν μάλλον γενική μόρφωση και μόνο το υπόλοιπο 20% έχουν επαγγελματική μόρφωση ή πανεπιστημιακό πτυχίο. Περίπου 70% είναι ηλικίες κάτω των 30 ετών, ενώ οι γυναίκες είναι κάτω του 30%. Αυτή είναι λοιπόν η αφετηρία και η κατάσταση που έχουμε ε, όταν ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ένταξή του στην αγορά εργασία. Τι σημαίνει αυτό για τη στρατηγική. Ε, η αγορά εργασία είναι καλά δομημένη στη Γερμανία και μπορεί να καταφέρει την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Επειδή δεν έχουν τυπικά προσόντα, για μας αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε τι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι και όχι να αναγνωρίσουμε τυπικά προσόντα γιατί συχνά δεν έχουν. Αλλά το να ε, καταλάβει τι δεξιότητε έχουν και τι προσόντα δεν υπάρχουν τέτοιε μέθοδοι και τέτοιε διαδικασίε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον όχι για τόσου πολλού ανθρώπου. Πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις κλίμακες και τι αυτές σημαίνουν. Δηλαδή δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα περιορισμένο ή ένας αριθμός που ε, μπορεί να περιοριστεί σε μια συγκεκριμένη επικράτεια, ας πούμε, μικρή. Ακριβώς λοιπόν, επειδή δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι τυπικά προσόντα, αλλά και επειδή είναι και τόσο νέοι, δικός μας στόχος είναι όσο γίνεται να τους ε, προσφέρουμε πλήρη κατάρτιση και εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι έχουν δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα, ακόμα και αν έχουν τα τυπικά προσόντα. Και θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά. Δηλαδή, αν βγούμε στην ενταξη αγορά εργασία, θέλουμε αυτό να συνδυαστεί με την εκμάθηση της γλώσσας, με την ε, έναρξη εργασίας και με ε, παροχή προσόντων και δεξιοτήτων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα ποτάρουμε στο να μην γίνουν οι σημερινοί πρόσφυγε ή οι αυριανοί μακροχρόνια άνεργοι. Γνωρίζουμε ανέκαθεν ναι, ότι στην πρώτη πενταετία μπορούμε να ενσωματώσουμε το πολύ πολύ τους μισούς. Αυτό είναι εμπειρία του παρελθόντος και θα πρέπει να βελτιωθούμε. Επίσης, άλλος στόχος. Να μην υπάρχει διακρίση ε, ε, εις βάρος των τόπιων, είτε αυτή είναι ε, Γερμανοί είτε είναι πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε πόσο τεταμένο είναι το κλίμα και δεν θέλουμε να οξυνθεί. Και υπάρχουν ε, ήδη προβλήματα ε, στην αγορά εργασίας που δεν θα πρέπει να παραμεληθούν. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα περίκοπες. Δεν αποκλείονται κάποιες συγκρούσεις και κάποιοι ανταγωνισμοί, αλλά αυτό αυτές κατά την άποψή μας ε, αφορούν μόνο τους ανειδίκευτους. Και τουλάχιστον στη Γερμανία ένα έκτακτο πρόγραμμα για πρόσφυγες δεν πρόκειται να ε, δημιουργηθεί διότι υπάρχουν ήδη εργαλεία και μέσα που προσφέρονται και μπορούν να αξιοποιηθούν για να ε, αποδώσει η προσπάθεια αυτή θα πρέπει βέβαια σε νέα κλίμακα να ενταχθούν, να προσαρμοστούν, αλλά όχι νέα εργαλεία. Τι κάνει λοιπόν η υπηρεσία εργασίας στη Γερμανία. Ακούσαμε το παράδειγμα από τη Σουηδία. Ε, έχουμε μια διαδικασία που ξεκινάει πολύ νωρίς ε, για να καταγράψουμε τα προσόντα και τις δεξιότητες εκείνων που έχουν καλές προοπτικές να παραμένουν στη χώρα και γίνεται μια πρώτη συνέντευξη σχετικά νωρί όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλέ πιθανότητε ένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασία. Ε, αυτή την ε, φιλοδοξία έχουμε. Δουλειά μπορεί κανείς να βρει στη Γερμανία ήδη μετά από τρεις μήνες. Ε, έτσι έχει το νομικό πλαίσιο. Και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό τον έλεγχο, του screening και το profiling ήδη από την αρχή, από τη στιγμή που κάποιος υποβάλλει αίτηση για εύρης εργασίας. Σας είπα το μοντέλο. Θέλουμε να συνδυαστεί ε, η εκμάθηση της γλώσσας, η εκμάθηση των δεξιοτήτων και η έβρεση εργασίας. Έχει αρχίσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα σύνδεση όλων αυτών με την παραγωγή και τις παραγωγικές διαδικασίες και τα προϊόντα. Έχουμε ήδη ειδικέ προσφορές για νέους πρόσφυγες αλλά και για γυναίκες. Τα προγράμματα ήδη έχουν δεσπιστεί και θα πρέπει να προσαρμόσουμε και το νομικό μας πλαίσιο για τις δυνατότητες στήριξης οικονομικής, για παράδειγμα. Κανονικά θεωρούμε ότι όταν κάποιος έχει ε, αποφοιτήσει από το σχολείο αλλά δεν έχει επαγγελματική κατάρτιση, ε, μόλις τελειώσει το σχολείο ε, υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθεί και να εκπαιδευτεί. Υπάρχει ένα ανώτατο ηλικιακό όριο σε αυτό, γιατί πρέπει να είναι κοντά στο σχολείο. Τώρα οι πρόσφυγες είναι ε, στην ηλικία λίγο μεγαλύτερη, αλλά επί της ουσίας πληρούν αυτά τα προσόντα και αντιστοιχεί η κατάστασή τους στην προηγούμενη ε, που σας ανέφερα, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο αυξήσαμε το προσωπικό μας αλλά και τους οικονομικούς μας πόρους τον προϋπολογισμό για να ε, χρηματοδοτήσουμε αυτό το επιπλέον ε, έργο και το φόρτο και επίσης επενδύουμε πάρα πολύ ε, στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και των συνεργατών μας για διαπολιτισμική αυτή η πραγματικότητα γιατί πολλούς είναι μια πολύ καινούρια εμπειρία και χρειάζεται να τη μάθεις και αυτή. Δηλαδή δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι μια διαδικασία στάνταρ σαν αυτή που γνωρίζω μέχρι σήμερα. Η υποστήριξη της ε, παροχής συμβουλών ε, από τον Απρίλιο θα διαθέσουμε μία τηλεφωνική γραμμή διερμηνής και ε, ε, βίντεο, τηλεδιασκέψεις και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με βίντεο. Χρησιμοποιούμε και τα νέα media. Έχουμε μία ιστοσελίδα υποδοχής, landing page και μία εφαρμογή που λέγεται άφηξη για την υποδοχή, την πρώτη επαφή και έχουμε κάποιες γλώσσες τις οποίες ενημερώνουμε ε, για τις δυνατότητες και θα ε, αυξηθούν αυτές οι γλώσσες, θα προσθεθούν άλλες 7. Αυτά. Είχα να σας πω και με χαρά περιμένω τις ερωτήσεις σας. Thank you, Mr. Uh, next Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μίλλερ. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Ντενί Αβό, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ερυθρό Σταυρό, την Ευρωπαϊκή Έδρα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Ερυθρού Σταυρού. Έχετε το λόγο κύριε Αβό. Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στην σημερινή ακρόαση. Εμείς εκπροσωπούμε τις ε, του 28 ερυθρούς σταυρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και τον Νορβηγικό Ερθρικό Σταυρό και τη Διεθνή Ένωση Ερυθρού Σταυρού. Θα γνωρίζετε ότι ο Ερυθρός Σταυρός αποτελεί ένα κίνημα το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει διάφορες καταστροφές και έκτακτες καταστάσεις, αλλά παρέχουμε επίσης και υπηρεσίες σε τοπικές κοινότητες, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 250.000 άτομα εργάζονται και πάνω από ένα εκατομμύριο θελοντές. Όλο και περισσότεροι πρόσφυγες πρόσφυγες φτάνουν ή περνάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως ο Ερυθρός Σταυρός και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχουν έντονη παρουσία αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο. Προσπαθούν να αποκριθούν στις ανάγκες των προσφύγων χωρίς καμία διάκριση και προσπαθώντας να προστατεύσουν το διεθνές καθεστώ του. 600.000 πρόσφυγες έχουν ήδη φτάσει μέχρι το Φεβρουάριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ένταξή τους. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σαφώς υπέρ της όλης εργασίας προβλέπεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχοντας μια συγκεκριμένη εμπειρία εργαζόμενη με και για τους πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να επικεντρωθώ στα επόμενα τρία σημεία και να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το τι μπορούμε να κάνουμε κάνουμε σε εθνικό επίπεδο και ποιε υπηρεσίε μπορούμε να παράσχουμε. Οι απαραίτητε καταρχά προποθέσει προκειμένου οι πρόσφυγε όντω να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Δεύτερον, να καταφέρουμε να προωθήσουμε επιπλέον υπηρεσίε ενσωμάτωση όχι μόνο των ίδιων των προσφύγων αλλά και των οικογενειών του και να πετύχουμε επομένω την επανένωση των οικογενειών και τρίτον να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία και τη διακριτική μεταχείριση. Πρώτον λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά εργασία για του πρόσφυγε και του ετούτε άσυλο ήδη από πάρα πολύ νωρί. Το να έχει κανεί μία εργασία πραγματικά διευκολύνει την κοινωνική του ένταξη, την κοινωνική του ενσωμάτωση και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει και αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση και στέγασης. Ωστόσο, Άρα πολλές προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα να πληρούνται προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των προσφύγων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες πολιτικές και πρακτικές που μπορούν πραγματικά να προωθήσουν την αποτελεσματική αυτή ενσωμάτωση του πρόσφυγα στην αγορά εργασία, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ιδιάζουσα κατάστασή του. Πάρα πολλοί πρόσφυγες, α μην το ξεχνάμε, έχουν περάσει από τραυματικές εμπειρίες, από τραγικές αντικσότητες προτού φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτού ασχοληθούμε λοιπόν με την ένταξη στην αγορά εργασία αυτή καθεαυτή, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ιδιαίτερε ανάγκε του. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προωθήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, προκειμένου όλα τα κράτη-μέλη να έχουν κοινά πρότυπα για την αγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πιστοποιητικών και άλλη σχετική εμπειρία των προσφύγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να δούμε τα λεγόμενα soft skills, ή δεξιότητε, όπω για παράδειγμα πρώτερη επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών. Προφανώ αυτά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ένταξη στην αγορά εργασία. Ξέρετε ότι στη Δανία υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα πρόγραμμα από τον εκεί Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να ή περνάνε από κάποια προγράμματα κατάρτισης και αναγνώρισης προσόντων οι πρόσφυγε προτού φύγουν από τα κέντρα υποδοχής. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουν περισσότερες πιθανότητες να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Θέλοντας επίση να ενισχύσουμε τι δεξιότητε των προσφύγων, θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Αυτές οι νέες δεξιότητες και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν θα πρέπει να προβλέπονται μόνο για τα παιδιά των προσφύγων. Επίσης, η απουσία των απαραίτητων κοινωνικών, οικογενειακών ή επαγγελματικών δικτύων καταστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη για τους πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Αντίθετα, οι πρόσφυγες εκείνοι οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι σε δίκτυα μπορούν να ενσωματωθούν πολύ πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού καθοδήγησης. Για παράδειγμα, ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός ήδη από το 2000 έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Επαγγελματικό Σχέδιο για τους Πρόσφυγες με απότερο στόχο να προσδώσει νέε δεξιότητε ή αναγνώριση φυσταμένων δεξιοτήτων στου πρόσφυγες και από την άλλη να του δώσει καλύτερε ευκαιρίε πρόσβαση στην αγορά εργασία. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται για μικρά πιλωτικά προγράμματα. Μόνο και μόνο το 2014 100.000 πρόσφυγες συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 31.000 από τα άτομα αυτά ήταν πρόσφυγες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης οι πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες όπως οι υγειονομικές υπηρεσίες ή οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πάλι από τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να υποστηρίζει κανείς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά να, υπάρχει, να υπάρχουν και τα απαραίτητα συστήματα υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορεί ο πρόσφυγας να έχει πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικέ υπηρεσίες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σχετική αναφορά όσον αφορά τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και προβλέπει ότι θα πρέπει και τα δικαιώματα αυτά να προβλέπονται για τους πρόσφυγες. Όσον αφορά τον Ερυθρό Σταυρό, ξέρετε ότι η εθελοντική εργασία συμβάλλει πάρα πολύ στην ομαλή ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν μέσω του θελοντισμού δεξιότητες, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια κατά την εργασία την οποία πρόκειται να βρούνε. Πέρα από αυτό, πέρα από την ενσωμάτωση στην αγορά εργασία, υπάρχουν και άλλα μέτρα υποστήριξη στην κοινωνία. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επανένωση των οικογενειών. Η ε, συνεχή, ε, θέλετε, ανησυχία, ένα συνεχέ άγχο για ένα πρόσφυγα, ο οποίο έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να επανενωθεί με την οικογένειά του. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, ο πρόσφυγα γίνεται όλο και πιο ευάλωτο. Η επανένωση λοιπόν με την οικογένεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, προκειμένου οι πρόσφυγε να γνωρίζουν, να ξέρουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν να ενσωματώνονται ομαλά στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η ε, Ευρωπαϊκοί Ερυθροί Σταυροί που βρίσκονται στι διάφορε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια την οικογενειακή επανένωση, δίνοντα νομικέ συμβουλέ προ του πρόσφυγε, καλύπτοντα πολλέ φορέ τι ταξιδιωτικέ δαπάνε των μελών τη οικογένειά του, προκειμένου να έρθουν και να επανενωθούν με τον πρόσφυγα που έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, έχουμε ομάδε δικηγόρων, οι οποίε συμβάλλουν στο να επιτευχθεί η οικογενειακή επανένωση των προσφύγων. Βασιζόμενοι λοιπόν σε εμπειρίε αυτέ, θεωρούμε ότι περισσότερα πράγματα θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταρριφθούν τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οικογενειακή επανένωση, όπως οι διοικητικές διαδικασίες, τα υψηλά ταξιδιωτικά κόστη, αλλά πολλέ φορέ και οι πολύ αυστηροί κανόνες όσον αφορά την παροχή θεώρησης, ταξιωτικής θεώρησης. Όσο καθυστερεί η οικογενειακή επανένωση, τόσο επιδεινώνεται η ζωή του πρόσφυγα. Υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν κάποιου περιορισμούς όσον αφορά το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης. Εμείς ακράταντα πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί εδώ να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, λέγοντα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προασπιστεί το δικαίωμα αυτό στην οικογενειακή ζωή και ότι αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για την ομαλή ενσωμάτωση των προσφύγων στι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Τέλο, υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν ξενοφοβία, ρατσισμό, διακριτική μεταχείριση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε εδώ πέρα να συνειδητοποιήσουμε ποιε είναι οι μακροπρόθεσμε ευκαιρίε που προσφέρει η προσφυγική κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τονίσει την κοινωνική, τη θετική συμβολή των προσφύγων σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Από το 2014 και μετά ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί να προωθήσει την θετική ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μέσω της εκστρατείας ότι κανένα ανθρώπινο όν δεν μπορεί να θεωρείται παράνομο. Ολοκληρώντας, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εξαιτία της μεγάλης αυτής έλευσης των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθίστανται όλο και πιο έντονε οι ανάγκε των προσφύγων αυτών, προκειμένου να καταφέρουν να ενταχθούν στι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Άρα, χρειαζόμαστε μέτρα όχι μόνο για την ένταξη στην αγορά εργασία, αλλά και επιπλέον συνοδευτικά μέτρα και υπηρεσίε, σαν αυτά τα οποία ανέφερε. Οικογενειακή επανένωση, δηλαδή πρόσβαση στι κοινωνικέ ε, υπηρεσίε, κοινωνικονομική υποστήριξη, ε, παροχή νομικών συμβουλών και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν προγράμματα για την ομαλή ενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά εργασία και γενικότερα σε ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Η ενσωμάτωση ένταξη είναι μια μακρόπνοη διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια τη άφηξη του πρόσφυγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προωθήσετε λοιπόν πολιτικέ οι οποίε θα συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων. Από κοινού όλοι πρέπει να εργαστούμε προκειμένου η ένταξη αυτή να αποτελέσει μια πραγματική λύση για τη ζωή των προσφύγων. Για άλλη μια φορά να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα και με διάθεσή σα για περαιτέρω πληροφορίε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ναι. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν εύκολε και γρήγορε λύσει. Θα ήθελα να καλωσορίσω και του υπόλοιπου προσκεκλημένου που έχουμε εδώ. 30 διοικητικού υπαλλήλου ε, του Νομαρχιακού Συμβουλίου τη Ακυτένη ε, Σαρόντ και Πουατού. Καλώ ήρθατε λοιπόν. Σα καλωσορίζω. Πού είσαστε καθισμένοι. Ναι, εντάξει, έχουμε και 11 μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου. Εσείς είστε εδώ. Πολύ ωραία. Η Ευρωπαϊκή, η Νορβηγία βρίσκεται στα νότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλες τις τοποθετήσεις μέχρι τώρα και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Αμπουμπακάρ Σουμαούρο ο οποίος εκπροσωπεί την, ε, το Συνδικάτο Unione Sindacale την και είναι αρμόδιος για θέματα μετανάστευση από την Ιταλία, ο κύριος Σουμαγόρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι μέλος ε, του συνδικαλιστικού προεδρίου σε εθνικό επίπεδο της Ένωσής μας, αλλά ταυτόχρονα και της Ένωσης, Διεθνούς Ένωσης για τους ε, μετανάστες, πρόσφυγες και ανθρώπους που δεν έχουν ε, χαρτιά διαμονής. Έχουμε παρουσία σε πολλές χώρες, τρεις ευρωπαϊκές, άλλες τρεις στην Αφρική. Και το να μιλούμε σήμερα για τους ε, πρόσφυγες στην αγορά εργασίας, το να μιλούμε για την κοινωνική ενσωμάτωση, συνιστά καταρχάς μια προσπάθεια να καταλάβουμε το θέμα στο εύρος του και το να πούμε στους ε, πρόσφυγες. Ε, έχω μια παρουσίαση και γι' αυτό θα ήθελα. Και να πούμε λοιπόν στους πρόσφυγες καταρχάς, το να μιλήσουμε μάλλον για τους πρόσφυγες καταρχάς σημαίνει αναφορά στα κείμενα των συμβάσεων των σχετικών με τους πρόσφυγες τα οποία περιγράφεται ως πρόσφυγας ως πρόσωπο παρένθεση ανθρώπινο όν που βρίσκεται σε χώρα εκτός εκείνης της οποίας έχει την ηθαγένεια ή την συνήθη διαμονή του, ε, λόγω διώξεων ή φόβου διώξεων που στηρίζονται στο οφείλο στην φυλή, συγγνώμη, τη θρησκεία, την ηθαγένεια, την υπαγωγή σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή τις πολιτικές του απόψεις. 60 εκατομμύρια πρόσφυγες στον κόσμο υπάρχουν από ό,τι μας λέει η τις πολιτικες του αποψεις 60 εκατομμυρια προσφυγες στον κοσμο υπαρχουν οπως μας λεει η πατιαρμοστια των Ηνωμένων Εθνών. 9 εκ των 10 αυτών ζουν σε, οικονομίες, σε χώρες με οικονομία λιγότερο ανεπτυγμένη αυτής από την οποία προέρχονται. Δεν ζουν δηλαδή ε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει εισβολή η σύμβαση, πολύ σημαντική σύμβαση, πρέπει να διαφυλαχθεί. Είναι πολύ σημαντική όμως η περιγραφή του όρου του πρόσφυγα με δεδομένες τις εξελίξεις, τις κοινωνικές και γεωπολιτικές της εποχής μας. Ο ορισμός λοιπόν αυτών, αυτός είναι ανεπαρκής. Για να αντιληφθούμε τους λόγους που οδηγούν στη φυγή, που προξενούν θανάτους που έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης σε νεκροταφεία είναι πάνω απ' όλα ζητήματα ανθρωπιάς και προσέγγισης. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στις τρεις διαστάσεις της προσέγγισης που είναι πρώτον η αντιμετώπιση κατεπίγουσας ανάγκης, αυτό που λέγεται μεταναστευτική κρίση, μια διάσταση που σημαίνει πως έχουμε μπροστά μας μια κατάσταση που απαιτεί κατεπίγουσα παρέμβαση, Μια κατάσταση που έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα στην πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 2015-2016 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια κατάσταση κατεπίγουσα, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς ορθολογική προσέγγιση, που σημαίνει απλώς τραβάω λεφτά από το ταμείο. Πολλές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όχι όλες, αλλά πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν καταστεί ειδικοί στην υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που χρειάζονται ενσωμάτωση. Δεύτερη προσέγγιση είναι η φιλανθρωπική προσέγγιση βλέπει ότι πρόκειται για θέμα καταρχά ηθικό, για θέμα δεοντολογίας το να υποδεχθεί κανείς του πρόσφυγες. Και έτσι πολλοί ε, τη χάνουν αυτής της υποδοχής. Η τρίτη προσέγγιση είναι η διαρθρωτική προσέγγιση, από την οποία θα ήθελα να δώσω κάποια παραδείγματα. Φερρυπίν το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών 2013 20 εκατομμύρια άτομα ε, εγκατέλειψαν τις αιστείες τους λόγω των κλιματικών αλλαγών. Δεύτερο στοιχείο αυτής της διαρθρωτικής ε, ε, προσέγγισης είναι αυτοί οι οποίοι λόγω ένοπλων συγκρούσεων εγκαταλείπουν τις αιστείες τους και αυτό είναι ένας από τους κύριους λόγους που οδηγούν κάποιον να εγκαταλείψει τη χώρα του. Και ένα τρίτο στοιχείο, αυτό το οποίο σχετίζεται με την οικονομία του πολέμου, ή καλύτερα τον οικονομικό πόλεμο. Οικονομικό πόλεμο ο οποίος οφείλεται σε πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες, στις οποίες σημειώνεται σημαντική οικονομική ανάπτυξη, 4,5% φερρυπίν για την υποσαχάρη Αφρική, με ταυτόχρονη όμως διάχυτη και πολύ διαδεδομένη φτώχεια, οφειλόμενη στα μέτρα που έχει επιβάλει το Διεθνέ Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα στι χώρε αυτέ. Το να μιλούμε λοιπόν για πρόσφυγε και αγορά εργασία με βάση την οδηγία 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τους όρους υπό τους οποίους εξασφαλίζεται η, προσφορά, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον ετούντα το άσυλο με βάση το εθνικό τους δίκαιο και με εγγύηση της ε, αποτελεσματικής πρόσβασης για τον ετούντα το άσυλο. Δηλαδή σε αυτή τη διάσταση έχουμε 28 κράτη-μέλη με κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο διαφορετικό το καθένα, δηλαδή διαφορετικά μέτρα πρόσβαση στην αγορά εργασίας για το κάθε ένα από τα 28 κράτη και αν δεν υπάρχει αυτή η διάσταση, αυτή η φωτογραφία σας δείχνει τι συμβαίνει, πρόκειται για τους εργαζόμενους στον χώρο της ε, γεωργίας που ζουν σε αυτές τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Βλέπετε τις, ε, τα ρούχα αυτά, τα απλωμένα, τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων. Αυτή είναι σκουπιδότοπος, τα παπούτσια. Πρόκειται για σκλάβους αυτής της νέας ε, χιλιετίας. Αυτή είναι η κουζίνα τους που βλέπετε. Εμείς για να αντιδράσουμε και να δράσουμε έχουμε ιδρύσει ως συνδικαλιστικό σωματείο ένα γραφείο ε, όπου καλωσορίζουμε και προσπαθούμε να προσφέρουμε πληροφορίες στους ανθρώπους αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι για να μιλήσουμε για αγορά εργασίας σημαίνει, ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση και αυτό σημαίνει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε τους όρους ε, πρόσβασης με αξιοπρέπεια για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και με ισότιμα δικαιώματα. Και για να ολοκληρώσω κάποιες προτάσεις που αφορούν την κοινωνική κινητικότητα και τη δυνατότητα της εγκατάστασης, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα που προβλέπει η ε, σύμβαση του Δουβλίνου, η συνθήκη του Δουβλίνου. Επίσης έχουμε την πρόσβαση στην κατάρτιση και την αναγνώριση των ε, τίτλων σπουδών, γιατί φτάνει κανείς σε μια χώρα, δεν μιλάει τη, γλώσσα της χώρας αυτής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην έχει κάποιες άλλες βασικές γνώσεις. Υπάρχει όμως το ζήτημα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών. Πρόβλημα επίσης αποτελεί η εναρμόνιση των διάφορων ε, πόρων που αφορούν ε, την υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων. Ο αγώνας κατά της ε, εκμετάλλευσης και της δουλείας, η νομιμοποίηση εκείνων που ζουν ήδη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεργασία, ο συντονισμός μεταξύ τοπικών και άλλων φορέων κοινωνικο-οικονομικών, η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κανόνων πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για να ολοκληρώσω το μόνο που μπορώ να παραθέσω είναι η φράση αυτή το μεγαλύτερο για μένα και πιο πολύτιμο ιδεώδες ήταν το ιδεώδες μιας ελεύθερης κοινωνίας, μιας δημοκρατικής κοινωνίας στην οποία όλοι θα μπορούσαν να ζήσουν σε αρμονία με ίσες ευκαιρίες. Λόγια του Νέλσον Αμαντέλα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σωμαχώρο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λέν Βεράστ, Γενική Διευθύντρια της Φλαμανδικής Υπηρεσίας Ενταξής στο Βέλγιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο today. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να κοιτάξω λίγο την παρουσίαση αν λειτουργούν τα συστήματα. Μάλιστα. Πάμε. Ε, ε, εργασία ίσον ένταξη ίσον εργασία. Αυτή είναι η βασική μας ε, φιλοσοφία στην υπηρεσία μας. Και τι σημαίνει αυτό. Τρεις βασικές αρχές που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε πρόσφυγες και σε όλα τα έργα και τα projects που κάνουμε με τους ε, εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η εργασία καταρχάς είναι βασικός παράγον για την επιτυχία σου. Δίνει εισόδημα, ταυτότητα και ρόλο στην κοινωνία η εργασία σε κάνει να έρχεσαι σε επαφή με άλλους ε, πολίτες, να μαθαίνεις καλύτερα τη γλώσσα και να βλέπεις πώς λειτουργεί μια κοινωνία. Δεύτερη αρχή. Ο πρόσφυγας δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα η λέξη πρόσφυγας και το καθεστώς είναι νομικό κατασκεύασμα και φέρει μαζί του κάποια δικαιώματα και κάθε, κάθε, κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά πάνω απ' όλα κάθε πρόσφυγας είναι άτομο με τη δική του ιστορία, με τη, δική του εμπειρία, με τις δικές του δεξιότητες, με τις δικές του ικανότητες να μαθαίνει. Και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη ε, αρχή μας ότι θα πρέπει να είναι κομμένη και ραμμένη κάθε δουλειά στα μέτρα του ενδιαφερομένου. Το πρόσωπο μας ενδιαφέρει, το άτομο και οι δεξιότητές του. Και αυτή είναι η αφετηρία και αυτό είναι και το κέντρο. Ε, είμαστε πάρα πολύ εστιασμένοι στην προσωπική συνέντευξη. Η φλαμανδική κυβέρνηση αναγνωρίζει τις βασικές αρχές πολιτική πολιτικής των προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά μεταφράζονται σε μια πολιτική ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών με μια μόνιμη διάδραση μεταναστών και κοινωνίας. Είναι διπλής κατεύθυνση αυτός ο δρόμο. Έχουμε στρατηγικούς στόχους από τη φλαμαδική κυβέρνηση και η υπηρεσία μας συντονίζει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται. Και μέσα σε αυτή την πολιτική κάθε υπουργό αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για να ελοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι. Γενικές πρωτοβολίες, ε, αν είναι δυνατό, και ειδικά μέτρα, αν είναι απαραίτητο. Η ε, τοπική αυτοδιοίκηση επίσης ε, ασχολείται με αυτά τα θέματα, οι μεγάλες πόλεις καταλαβαίνετε ότι έχουν άλλα προβλήματα από ότι ε, κάποια μικρά χωριά ή κοινότητες στην Ήπεθρο. Τι δίνουμε, τι προσφέρουμε στους ε, νεοαφιχθέντες. Ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης στην κοινωνία που λέγεται Inburgering στα Ολλανδικά και είναι ένα πρόγραμμα αγωγής του πολίτου και εκμάθησης της γλώσσας. 4.700 ευρώ επενδύει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα και είναι δωρεάν για τους ε, συμμετέχοντες. Εκείνοι όμως που γράφονται στο πρόγραμμα αυτό να αναμένεται και να το τελειώσουν και να αποφυτίσουν. Επίσης, επιδοτεί η κυβέρνηση ε, μία ε, οργάνωση συμμετοχής και ένταξή τους στην κοινωνία έτσι ώστε γίνεται ε, δουλειά και υπάρχει και ξεχωριστή υπηρεσία οργανισμό τη κυβέρνηση για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Υποστηρίζουμε τι δημόσιε υπηρεσίε, του ΟΤΑ, την κοινωνία των πολιτών στη συνεργασία με του μετανάστε. Ε, με ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση για τα δικαιώματα στέγασης, τις νομικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, διερμηνία κτλ. Επίσης συλλέγουμε και μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές με περισσότερη συμμετοχή τους στην κοινωνία, ε, με διάφορα κοινά προγράμματα. Αφιερώνουμε την περισσότερη δραστηριότητά μας, 18.000 προγράμματα κάθε χρόνο. Ε, θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να σταθούν στα πόδια τους, να μάθουν Ολλανδικά, να βρουν δουλειά και να λειτουργούν στην κοινωνία πάντα με βάση τον άνθρωπο και τη μεμονωμένη περίπτωση. Όποιος φτάνει για ε, πρώτη φορά στη Φλάνδρα ε, πρέπει να χαράσει ένα σχέδιο, πώς θα πάρει τη ζωή του στα χέρια του και θα αναλάβει τις ευθύνες του. Και με αρχές και προδιαγραφές που συζητούμε, οι οποίες είναι βασικές για την κοινωνία μας και έτσι μαθαίνουν και τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις και τι εστί να ζεις στη Φλάνδρα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ε, τον προετοιμάζουμε επίσης και την ένταξή του στην αγορά εργασία. Η εξελόγηση του προγράμματος μας δείχνει ότι οι περισσότεροι αφιχθέντες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την υπηρεσία, παρόλο που γνωρίζουν ότι είναι και υποχρεωτικοί και χρειάζεται να κάνουν ήδη μεγάλη προσπάθεια. Ε, ε, κάνουμε ε, προγράμματα άσκησης και μαθητείας στις εταιρείες και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και όλα αυτά που μαθαίνουν κατά τη διάρκεια της μαθητείας μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτή τη στιγμή εργοδοτηθούν. Με βάση την εμπειρία μας θα κάναμε τις εξή πέντε συστάσεις. Πρώτον, και ακούστηκε και προηγουμένω αυτό, πρόορη, η έγκαιρη ε, παρέμβαση είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει πολύ γρήγορα να πάρουμε στα χέρια μας ε, έναν ελτούντα άσυλο και ταυτόχρονα ελέγχοντας το πρόγραμμα ε, και αυτό είναι υποχρεωτικό για τους πρόσφυγες που έχουν αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα. Η ένταξη είναι αμοιβαίως επωφελής και για την κοινωνία και για εκείνο που φτάνει σε μια κοινωνία. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα στοχευμένα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του καθενός. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα για όλους. Αυτό είναι εγγύηση αποτυχίας και αποθαρρύνει και τον κόσμο και τον αποκαρδιώνει. Η ενσωμάτωση και ένταξη σε μια κοινωνία και σε μια αγορά εργασίας είναι περίπλοκη ε, υπόθεση και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες επιτυχίας. Ε, μπορεί να έχει ένα κοινό στόχο, αλλά χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση. Η συνεργασία μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου και οργανώσεων είναι εκ των όνου κάνευ. Μπορεί να σας φαίνεται λογικό, αλλά στην πράξη αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο. Η ένταξη πολύ συχνά ε, είναι κάτι που βλέπει κανείς από μία και μόνη σκοπιά. Επίσης, η γλώσσα είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για να μπορεί να ενταχθεί κάποιο στην κοινωνία. Η εκμάθηση της γλώσσας θα πρέπει να γίνεται όσο γίνεται πιο κοντά στην πρακτική, στην καθημερινή ζωή και μεταξύ αυτών και στην αγορά εργασία και στον χώρο εργασίας μάλλον. Η κάθε συζήτηση είναι η δυνατότητα και ευκαιρία να ε, χρησιμοποιήσει μια γλώσσα και να τη μάθεις. Για να μπορεί και ο πελάτης να ε, καταλάβει τι σημαίνει να μιλάει μια γλώσσα και τι ευεργετήματα θα έχει να μάθει. Και τέλος, η ενσωμάτωση και η ένταξη ε, χρειάζεται προσπάθεια και από την κοινωνία και από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και οι εταιρείε και οι κοινωνίες των πολιτών, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι πολίτες και οι ίδιοι μετανάστες. Είναι μια αμοιβαιότητα αυτή, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητή και ορατή. Πρέπει ο καθένας να καταβάλει κάποιο κόπο η επικοινωνία επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίζονται, να γκρεμίζουν τις προκαταλήψεις τους και να αρχίζουν να χτίζουν ένα κοινό μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Ο τελευταίος μας ομιλητής, ο κύριος Σχολεβίνσκι, ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και εκπροσωπεί τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όμως και τον κύριο Μπονιφάη, τον ε, εισηγητή σας, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας, της Επιτροπής σας, οι οποίοι ε, μας προσκάλεσαν σήμερα πρόσφυγες και σ' άσυλο στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και μας. Πρέπει να ισχύουν και για αυτούς διεθνή πρότυπα εργασίας και επομένως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ασχολείται ιδιαίτερα με την απασχόληση των προσφύγων αυτών. Βλέπουμε όλο και περισσότερο τη η διεθνής κοινότητα συντοποιεί ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή όχι μόνο να έχουμε μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και μια αναπτυξιακή αντιμετώπιση της κρίσης. Στη συνδιάσκεψη που κάναμε τον Ιούνιο του 2015 συζητήσαμε ακριβώς το ζήτημα αυτό και τον Νοέμβριο το Διοικητικό μας Συμβούλιο ανταποκρινόμενο στην, ε, στο τριμερές συμβούλιο του ILO θελήσαμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης από την προσφυγική κρίση και το τριμερές αυτό συμβούλιο θα συνεδριάσει και τον ερχόμενο μήνα όπου θα καλέσουμε τους εταίρους μας, διάφορες υπηρεσίες δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών, προφανώς την είπα τη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και άλλους όμως οργανισμούς, να συζητήσουν για το ζήτημα αυτό. Εμείς ως Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία για τους πρόσφυγες και αυτό αποτελεί μέρος του γενικότερου πλαισίου προστασίας τους. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με την ύπατη αρμοστία των ΗΕ προκειμένου να ασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή διαβίωση προσφύγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να έχουν λοιπόν οι πρόσφυγες πρόσβαση στην αγορά εργασίας και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουν και πρόσβαση σε δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό συνάδει με την νέα, το νέο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης του 2013, όπου λέγεται ότι η εξωπρεπής εργασία και η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελούν δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους και για τους πρόσφυγες. Ξέρουμε επίση ότι οι πρόσφυγες, οι ετούντε άσυλο και οι μετανάστε μπορούν να δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο και να συμβάλλουν πολύ σημαντικά στο σύνολο τη κοινωνία, φέρνοντα τη δική του συμπεριγνωμοσύνη, τα δικά του ταλέντα και τι δικέ του δεξιότητε. Αυτό ισχύει για τι χώρε προορισμού, για τι χώρε διέλευση και βέβαια μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των προσφύγων και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη δημογραφική κρίση σε διάφορε χώρε και τη μείωση του ενεργού πληθυσμού. Όπω έχει πει άλλωστε και ο Γενικό Διευθυντή μα, η υφιστάμενη προσφυγική κρίση είναι μια κρίση πολιτική, επιλογή πολιτική τελικά, που συμπεριλαμβάνει τόσο τα βαθύτερα αίτια της προσφυγικής κρίσης όσο και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τα αίτια αυτά. Δεν προκαλεί λοιπόν εντύπωση το γεγονός ότι με τις τόσο προσφύγων όσο και άλλων, όπως οικονομικών μεταναστών, επικεντρώνονται περισσότερο προς χώρες οι οποίες παρέχουν τις πιο ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, όπως η Γερμανία ή η Σουηδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε του θεσμού αγορά-εργασία, καθώ επίση και την ενημέρωση για την αγορά εργασία στι χώρε αυτέ, να έχουμε επίση καλύτερα δεδομένα, καλύτερη έρευνα και ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να καταφέρουμε να χαράξουμε τι κατάλληλε πολιτικέ και να υπάρχει επίση και η κατάλληλη γράμμιση πολιτικών και κατά την άποψή μα είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε την απαραίτητη ικανότητα των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, καθώ επίση και άλλοι εκπρόσωποι Τη κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν. Η βασική πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες, καθώς επίσης και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία και να αντιμετωπίσουμε του φόβου που έχουν οι πρόσφυγε αυτοί, καθότι βλέπουν ότι υπάρχει μια έντονη αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητά του αυτή να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Είναι πολύ σημαντικό επίση να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απαραίτητη χρηματοδότηση επίση. Τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου η γενικότερη ρητορική, η πολιτική ρητορική αυτή τη στιγμή να γίνεται πιο ενθαρρυντική. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον κατακαιρματισμό τη αγορά εργασία και να έχουμε ισότιμη μεταχείριση των προσφύγων σε όλου του οικονομικού τομεί. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα για την εργασία που κάνει η Διεθνή Οργάνωση εργασία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, στι χώρε εκείνε όπου οι προκλήσει ενσωμάτωση στην αγορά εργασία είναι πολύ μεγαλύτερε. Για παράδειγμα, στην ε, σχετική ανάλυση που κάναμε σε χώρες όπως η Ορδανία ή ο Λίβανος, ξέρετε δύο χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει πάρα πολλούς πρόσφυγες. Βλέπουμε λοιπόν στις χώρες αυτές ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική επίπτωση στην αγορά εργασίας από την έλευση των προσφύγων αυτών. Πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα εκμετάλλευση, επαγγελματική εκμετάλλευση των προσφύγων και πολλές φορές φτάνουμε ακόμα και σε καταναστική εργασία και μάλιστα ακόμα και σε καταναγκαστική παιδική εργασία. Και βέβαια αυτό είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα αρνητικό που κατ' επέκταση επηρεάζει και του υπόλοιπου εργαζομένου. Στην Τουρκία προσπαθούμε να δούμε πώ θα εφαρμοστεί η πρόσφατη νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων σε διάφορε καλλιέργειε, στον αγροτικό τομέα προσπαθούμε εδώ πέρα να δούμε κυρίω περιοχέ εκείνε τη Τουρκία που έχουν πάρα πολλού Σύριου πρόσφυγε. Να καταφέρουμε δηλαδή να έχουμε καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη κατάρτιση τόσο των προσφύγων όσο και των ε, υπευθύνων τη αγορά εργασία στι περιοχέ αυτέ τη Τουρκία. Κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύονται, θέλετε, και οι δύο πλευρέ και ενημερώνονται και οι δύο πλευρέ. Επίση, συνεργαζόμαστε στην Τουρκία με διάφορε υπηρεσίε απασχόληση, με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώ επίση και με του ε, Εργοδότε και του συνδικαλιστέ προκειμένου να έχουμε καλύτερη ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασία. Και στο σχέδιο αυτό υπάρχει και μια έντονη εκστρατεία ενημερωτική προκειμένου να περάσουν τα θετικά μηνύματα και να αλλάξει η στάση που αντιμετωπίζει ο κόσμο του πρόσφυγε, Να αναπτύξουν δηλαδή πιο θετικά αισθήματα προ αυτού. Το 2015 όντω φτάσανε πάρα πολλοί πρόσφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βέβαια δεν φτάσαμε σε καμία περίπτωση τα υψηλά ποσοστά προσφύγων που έχουμε σε χώρες όπως η Τουρκία, η Ορδανία και ο Λίβανος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο όσον αφορά την πρόσβαση των ετούντων άσυλο και των προσφύγων στην αγορά εργασία, που εφαρμόζεται το πλαίσιο αυτό σε 25 τουλάχιστον κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμω να δούμε πώ εφαρμόζεται στην πράξη και το πλαίσιο αυτό. Το Νοέμβριο του 2015 οργανώσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία εκδήλωση όσον αφορά την ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί ενδιαφέρομενοι φορείς συμμετείχαν, προφανώς πολλοί ευρωβουλευτές παρουσίασαν τη χώρα τους ή τη στάση των πολιτικών τους κομμάτων, ιδίως στις χώρες διέλευσης και προορισμού. Είχαμε επίσης οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, η Business Europe, η Ευρωπαϊκή Στομοσπονδία συνδικάτων και μη κυβερνητικοί ε, οργανισμοί συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή θελήσαμε να περάσουμε κάποια σημαντικά μηνύματα στα οποία έχουν αναφερθεί ήδη κάποιοι προαλήσαντε. Η ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασία σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερκεράσουμε την έλλειψη ελληνική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω μετά το ξέσπασμα τη Συριακή κρίση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τη βάση γνώσεων που έχουμε, να αλλάξουμε τα μηνύματα τα οποία προωθούμε, να καταρρύψουμε μύθου, να καταρρύψουμε στερεότυπα και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού μπορεί να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα άλλο σημαντικό μήνυμα προσπαθήσαμε να περάσουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την τεράστια αυτή έλευση των προσφύγων, ιδίως προς τις ε, νότιες χώρες. Ακούσαμε το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία έχει την απαραίτητη υποδομή, άλλες χώρες όμως δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα και τις απαραίτητες υποδομές. Όπως είπαν και κάποιοι προαλήσαντες, η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας μπορεί να βοηθήσει τη γενικότερη ομαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία. Είπαν επίσης οι προηγούμενοι ομιλητές ότι όσο πιο νωρίς καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση του πρόσφυγα στην αγορά εργασίας, τόσο βελτιώνεται η αξιοπρέπεια της ζωής του και η γενικότερη καλύτερη διαβίωσή του. Και αυτό είναι πολύ πιο θετικό επίσης ακόμα και για το δημόσιο κορβανά. Θεωρούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι οργανισμοί των εργαζομένων και των εργοδοτών να συμβάλλουν και αυτοί στην ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας μέσω συγκεκριμένων συλλογικών διαπραγματεύσεων και προσπαθώντας να κατευνάσουν κάπως τους ενδιασμούς ή τις ανησυχίες που έχουν κάποιοι εργαζόμενοι ντόπιοι σε ορισμένε περιοχέ, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Επίση πρέπει να έχουμε κάποια συνοδευτικά μέτρα όπω ε, και υπηρεσίε διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των προσφύγων στον χώρο εργασία. Η συμμετοχή αυτή ενεργή των προσφύγων στην αγορά εργασία δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει παράλληλα να έχουμε και κάποια μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εργασιακή κινητικότητα. Επομένω, θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε πιο νόμιμες οδούς έλευσης προσφύγων και μεταναστών προς τις αγορές εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους οικονομικού κλάδους και σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων. Επίσης, οι μετανάστες δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται, θα πρέπει να μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους και να καταπολεμούμε επίσης κάθε μορφή διάκρισης, είτε απέναντι στους νόμιμους είτε απέναντι στους παράνομους μετανάστες. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ζήτημα των δεξιοτήτων των προσφύγων που θα πρέπει να αντιστοιχούν με τι ανάγκε αγορά-εργασία. αφού το κάλυψαν και άλλοι ομιλητέ. Και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε δικαλιστικέ οργανώσει, οργανώσει εργοδοτών και επιχειρήσει και ανάμεσα στι κυβερνήσει βέβαια. Στη Γερμανία πάλι έχουμε ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Ήδη από την συνεδρίαση του Νοεμβρίου μάθαμε ότι υπήρχε πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και του Υπουργείου Μετανάστευση. Ξέρετε ότι είναι αυτά τα δύο Υπουργεία τα οποία ασχολούνται περισσότερο με τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα και την ε, ενσωμάτωσή του στην αγορά εργασία. Τα δύο λοιπόν αυτά υπουργεία στη Γερμανία συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά με την εκεί υπηρεσία απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να εμπλέξουμε πέρα από του κυβερνητικού φορεί και του κοινωνικού εταίρου. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θέλει να υποστηρίξει τις προσπάθειες της δικής σας Επιτροπής και γενικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και τα ίδια τα κράτη-μέλη προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Και βέβαια θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ε, υποστήριξη και των όμορων κρατών εκείνων που των όμορων κρατών ε, των κρατών μάλλον που βρίσκονται πολύ κοντά στις χώρες εκείνες που έχουν ε, δεχθεί πολύ μεγάλα ποσοστά προσφύγων. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε παρατηρήσεις και ερωτήσεις από τους ε, συναδέλφους. Γιούτα Στάντρουκ πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θερμά. Πολύ σημαντικές και ενημερωτικές τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρατήρηση ότι πρέπει οι κανόνες να ισχύουν για όλους, είτε πρόκειται για Ευρωπαίους, είτε πρόκειται για πολίτες από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για ένα πεδίο έντασης που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουν ή να μάθουν εξ αρχής να ξαναμάθουν όλα αυτά τα οποία απαιτεί η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Και ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει με την πρόκληση οι κοινωνίες μας να γίνουν ανοιχτές στην ενσωμάτωση και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να ε, βοηθήσουμε ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τα αιτήματα των ε, προσφύγων. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι από πλευρά των κρατών μελών και των υπηρεσιών τους να έχουν μια υποστήριξη και παρακολούθηση όπως και οι πρόσφυγες. Ιδιαίτερα θέλω να αναφέρω ότι η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας με επιδοτούμενες θέσεις πρέπει να προωθηθεί όπως είπα, μέσω των επιδοτήσεων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κοιτάξουμε και το ζήτημα του πώ αντιδρούν εκείνοι οι οποίοι στην Ευρώπη είναι χρόνια άνεργοι. Γιατί πρέπει και εκεί να δούμε πώ θα δώσουμε κάποιες λύσεις. Δεν μπορούμε να του λησμονήσουμε, πρέπει και αυτούς να του βάλουμε μέσα στο ε, πλάνο. Και αυτό σημαίνει να προσφέρουμε θέσει εργασία σε όλου, είτε πρόκειται για τον ε, άνεργο, το μακροχρόνιο άνεργο ή τον προερχόμενο από μια άλλη χώρα του κόσμου. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ε, μέσα στην Ευρώπη μεγάλη ε, ανεργία. Άλλες όμως περιοχές έχουν, ε, έλεια, έχουν έλλειψη σε εργατικό δυναμικό και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα δώσουμε τις λύσεις σε αυτό που ονομάζουμε στην Γερμανία υποχρέωση διαμονής και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε εσείς κάποιες προτάσεις. Μετά ακούσαμε για μελέτες και έρευνες των σωματείων του Ερυθρού Σταυρού, ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, προτάσεις που στηρίζονται σε μακρά εμπειρία. Ερωτώ λοιπόν υπάρχει μια εντατική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις βέλτιστες πρακτικές, φερειπίν στην Ισπανία για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και, αντί πολύ σημαντικό, Διαβάσαμε στη μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ότι οι μετανάστες, που, οι άνθρωποι που προέρχονται από χώρες άλλης Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο σαν ε, σκλάβοι, ε, εργάζονται δηλαδή σε συνθήκες ε, σκλαβιάς χωρίς δικαιώματα, χωρίς καν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να δεχθούμε εμείς στην Ευρώπη. Υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη κατάχρηση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Και νομίζω ότι έχουν σύμφωνη τοποθέτηση όλοι ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μονάδες παροχής συμβουλών. Είναι απαραίτητο αυτό και υπάρχουν καλά παραδείγματα όπου θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Και πολλές άλλες ερωτήσεις θα είχα βέβαια, αλλά ήδη μερός, για να μην σας καθυστερήσω παραπάνω, ή αν έχω πάλι την ευκαιρία της υποβάλλω σε μια δεύτερη τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ, μια και είναι πολύ λίγοι οι συντονιστές εδώ. Δίνω το λόγο στον επόμενο κύριο Ντομίνικ Μαχτάν. Με συγχωρείτε, η κυρία Λάμπερτ πρώτα από τους πράσινους. Προηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις και βέβαια θέλω να επισημάνω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αρκετές πληροφορίες από ένα σχέδιο που λέγεται Equal που είχε παρακολουθήσει πριν από μερικά χρόνια τους πρόσφυγες και τα ζητήματα της κατάρτισης, της επαγγελματικής, της εκμάθησης γλωσσών, της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και διάφορα άλλα ζητήματα που δεν πρέπει να λησμονηθούν. Ιδιαίτερα θέλω εγώ να ρωτήσω σε σχέση με την αλληλεπίδραση άδεια παραμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, πόσο μπορεί η άδεια παραμονής να την επηρεάσει, Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κάποιος έχει μια επικουρική ε, προστασία με μια άδεια παραμονής που ξεκινάει σε ε, μονοετή βάση και μετά γίνεται διετής και ούτω καθεξής, αν και αυτό βέβαια δεν ε, προσφέρει πολλές δεν απαλλάσσει από τη γραφειοκρατία των αντίων μάλλον. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι είδου πρόσβαση μπορεί να έχει κάποιο, ο οποίο ξεκινάει με μια μονοετία μονοετή άδεια παραμονή. Μήπω είναι αυτό τελικά φραγμό και εμπόδιο. Και επίση αξιολόγηση ε, δεξιοτήτων των ε, νεοαφιχθέντων, γιατί ασφαλώς δεν θα έχουν μαζί τους ε, οι άνθρωποι αυτοί τα πτυχία τους. Ξέρουμε ότι η πρόσβαση σε ε, έγγραφα ε, επίσημα από τη Συρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν μας εκπλήσει, αλλά πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και συστημικά πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα της αξιολόγησης των ε, προσόντων και δεξιοτήτων που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και ταυτόχρονα διευκολύνοντά του φυσικά, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση και ευχερέστερη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ κύριε Μαχτάντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ η συνάντησή μας, συνεδρίασή μας, κοινωνική ενσωμάτωση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, των προσφύγων είναι το θέμα της διασκεψιάς μας. Άκουσα τους πολύ καλούς ομιλητές και τους έξι, ε, αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση άκουγα να τοποθετούνται δηλαδή. Οι πρόσφυγες, η μετανάστευση αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη και δεν θα πρέπει να ε, στερηθούμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Δηλαδή έχει γίνει η Ευρώπη στοργή και προδέρμ. Ε, ρωτώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, αν είναι όλα τόσο καλά, τι την κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση. Τι καθόμαστε να συζητήσουμε το πρόβλημα αυτό. Γιατί προφανώς ούτε απλό είναι, ούτε προφανές αυτό που συζητούμε. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, δεν έχει γίνει διαφοροποίηση ε, για το αν πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες, εάν πρόκειται για οικονομικούς πρόσφυγες ή ακόμη και αν πρόκειται για τρομοκράτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις ε, γραμμές, ε, τις ε, ρότες της μετανάστευσης για να μπουν στην Ευρώπη. Ε, κάποιοι από εμά έπεσαν θύματα αυτών των τρομοκρατών μέσα στο 2015. Και είπε η κυρία Μακάριου νωρίτερα ότι οι πρόσφυγες έχουν χάσει τις ρίζες τους, η πρόεδρος. Με συγχωρείτε ένα λεπτό γιατί δεν ακούγεται η πολωνική mm. διερμηνία. Μπορούμε παρακαλώ Τώρα δουλεύει ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε. Κυρία Μακάρη, ε, η κυρία Μακάρη το επαναλαμβάνω, το είπε πολύ καλά. Έχουν ε, ξεριζωθεί, έχουν χάσει τις ρίζες τους, είναι δυστυχισμένοι μακριά από τις οικογένειές τους οι άνθρωποι αυτοί. Και φαντάζομαι ότι, ότι μόνος τους καημός και προσδοκία είναι η επιστροφή στις αιστείες τους. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρώπη λοιπόν είναι πάνω απ' όλα για μένα να τους βοηθήσει να επανέλθουν στις χώρες προελεύσεων έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβρούν το χαμόγελο και την ευτυχία τους. Μιλήσαμε επίσης για ενσωμάτωση, αλλά δεν μιλήσαμε για αφομοίωση. Όταν μιλούμε για ενσωμάτωση, και η κυρία Ακαρή ε, το παρέλαβε, ε, εννοούμε απαιτήσει και διαφύλαξη των χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένη κοινότητας. Η κυρία Ακαρή μιλάει για μια νέα κίνηση. Ναι, αλλά αυτή η νέα κίνηση δεν σημαίνει ενσωμάτωση, αλλά αποδοχή και ενστερνισμό των ηθών και εθήμων μιας κοινωνίας, όπως συνέβη στην, στις ΗΠΑ ή την Αυστραλία, χώρες των οποίων η οικοδόμηση δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Σημειώνω και λυπούμε. Άκουσα πολλές εκδικήσεις να εκφράζονται. Θέλω, πρέπει, θα οφείλατε. μάλιστα προσαρμοστούν και οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών. Δεν άκουσα πουθενά να εκφράζονται ευχαριστίες όμως. Δεν άκουσα ποτέ να λέει, να λέει ε, «Α, τι καλή η Ευρώπη που μας δέχεται και μας υποδέχεται». Φαντάζομαι ότι οι κάτοικοι της κολονίας στη Γερμανία θα έχουν μια διαφορετική θεώρηση αυτής της ε, έννοιας της υποδοχής και της γενναιοδορίας. Άκουσα και τον εκπρόσωπο της Γερμανίας να μιλάει. Όμως η Γερμανία είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Δεν είναι συγκρίσιμη με τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη. Η Γερμανία χρήζει εργατικού δυναμικού λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει. Αυτό δεν ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης και δι τη Γαλλία για την οποία σας πενθυμίζω έχουμε 6 εκατομμύρια ανέργους. Αυτά τα 6 εκατομμύρια άνεργοι της Γαλλίας ήδη αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα και εκφράζονται μέσα από ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό των μεγάλων ε, ε, πολυκατοικιών και συγκροτημάτων στα προάστια των ε, μεγαλού πόλεων, όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα ενσωμάτωσης και επίσης υπάρχουν, όπως υπόθηκε νωρίτερα, 28 συστήματα διαφορετικά ενσωμάτωσης. Άρα, εν τέλει και στο τέλος του λογαριασμού δεν βλέπω καμία δυνατότητα για ε, ενσωμάτωση και ούτε νομίζω ότι θα μπορούσατε να βρείτε τη λύση που αναζητάτε. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω και να επαναλάβω πως η μετανάστευση είναι μία τραγωδία. Πρώτα θύματα της μετανάστευσης είναι οι ίδιοι μετανάστες. Θάνατοι. Έγινε λόγος για τη Μεσόγειο που έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο. Ανεπαρκείς συνθήκες στέγης, εκμετάλλευση, μαφιόζικες οργανώσεις που καταχρώνται. Και θα σας ε, αναφέρω και πάλι κύριε Σουμαχώρο, είπατε πολύ σωστά ότι η μετανάστευση είναι η σύγχρονη δουλεία. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Υποδεχόμαστε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά τους υποδεχόμαστε, μάλλον τους υποδέχονται για να τους εκμεταλλευτούν. Ενώ θα έπρεπε να τους βοηθούμε να επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Και για να ολοκληρώσω συμπερασματικά, εδώ και μια μισή ώρα παρακολουθώ τις ομιλίες σας και μιλάτε σαν να μην υπάρχει λαό στην Ευρώπη, να μην υπάρχουν λαοί στην Ευρώπη. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη των ευρωπαϊκών λαών, γιατί να συμφωνήσουν οι λαοί της Ευρώπης με αυτό που αποφασίζετε εσείς. Δεν είναι προφανές και σας καλώ να το αναλογιστείτε. Και σας ευχαριστώ. Thank you, <coughs> Madame Κυρία Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει να πει πράγματα και λόγο για το θέμα αυτό και λυπάμαι που δεν σεβαστήκατε την καθιστική ατάξη εδώ και τη σειρά των πολιτικών ομάδων και δεν δώσατε ως οφείλατε το λόγο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όταν ήταν η ώρα του. Ελπίζω να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση. Βεβαίως είδαμε και ακούσαμε από όλους τους ομιλητές ότι η Ευρώπη παραμένει φάρος για όλους τους λαούς. και κυρίως χάρη στις αξίες που ενσαρκώνει και αντιπροσωπεύει και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε εύκολη ε, ξενοφοβία που πολύ γρήγορα μπορεί κανείς να πέσει σε αυτή σε αυτό το θέμα των μεταναστών. Θα ήθελα να χαιρετήσω τα όσα υπόθηκαν για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και το συνδέω με το προηγούμενο. Τα κράτη όντως έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Οι μήκοι όμως εκπροσωπούν την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών ακριβώς. Και αυτό είναι σημαντικό να έχει ρίζες στο λαό. Να μην είναι μια κινητοποίηση επιβεβλημένη άνωθεν, αλλά να είναι εξίσου ε, Και από την εμπειρία που έχω, από παραδείγματα επιτόπου, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή των ΜΚΟ στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Και θέλω πραγματικά να εξάρω το ρόλο τους. Δεν θα πετύχουμε εάν ε, ασκούμε μόνο εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές χωρίς τη συμμετοχή και ρήμην της κοινωνίας των πολιτών. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπε ε, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας για το τρίπτυχο που προωθούν από κοινού. Δηλαδή την εκμάθηση της γλώσσας, την ε, επαγγελματική κατάρτιση και την προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Συχνά ε, αυτούς τους, τους τρεις κρίκους της αλυσίδας τους υιοθετούμε διαδοχικά Κακός. Θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται και τα τρία. Ε, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ακριβώς αυτό το χρόνο για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τη Γερμανική Υπηρεσία Απασχόλησης τι γίνεται με την ειδική κατάρτιση των συνεργατών σας που είπατε ότι τους προετοιμάζετε για να ε, υποδέχονται ανθρώπους από διάφορους πολιτισμούς. Αυτή τη δυσκολία την αντιμετωπίζουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουμε υπηρεσίες ε, υποδοχής ανέργων, οι οργανισμούς έβρεσης εργασίας, αλλά που έχουν μια κατάρτιση και μια εκπαίδευση για τους ντόπιου. και δεν έχουν αυτή την οτροπία ε, του πολιτισμικού χαρακτήρα της υπόθεσης και ε, εξέπληξε αυτό που μας είπατε ότι υποδέχεστε ε, online σε 7 γλώσσες. Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ αυτό που είπατε για την κινητοποίηση των δικτύων. Τι βλέπω εγώ στην πράξη. Όντως ισχύει αυτό. Και η πρώτη κινητοποίηση ποια είναι. Όταν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά των μεταναστών δημιουργούνται δίκτυα για την ένταξή τους γύρω από τους μετανάστες αρχίζει λοιπόν από τη σχολική υποδοχή αυτή η προσπάθεια και επεκτείνεται. Εκεί όμως έχω ένα πρόβλημα το οποίο πάλι αντιμετωπίζω στην πράξη επιτόπου και θέλω να ρωτήσω πώς το έχουν λύσει οι ομιλητές μας και πώς το αισθάνονται και το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποια κέντρα υποδοχής που κινητοποιούν το σχολείο, τη ΜΚΟ, τα δίκτυα ολόκληρα. Στη συνέχεια καλούνται να αντιμετωπίσουν και την επαγγελματική ένταξη. Αλλά η επαγγελματική ένταξη δεν είναι εκεί που βρίσκεται το κέντρο υποδοχής. Δηλαδή γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες και μετά χρειάζεται και μια δεύτερη μετανάστευση, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, αλλά δεύτερη γεωγραφική μετακίνηση. Και θα πρέπει από την αρχή να στήσεις νέα δίκτυα ε, και όλη αυτή τη ζωή που είχαν χτίσει ήδη και όλο αυτό το περιβάλλον και για τα παιδιά και για τους γονείς στο νέο τόπο εργασίας. Και αυτή η νέα μετανάστευση, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες, αλλά στη δική μου χώρα δεν είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή χρειάζεται και πάλι από την αρχή να ανοίγει αυτό και χρειάζεται να προβληματίσει τους πολιτικούς. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια για να βελτιθεί η επικοινωνία με τα μίντια. Αυτά που βλέπω και ακούω από τα μίντια δεν είναι αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί. Και όσα κυκλοφορούν στα ΜΜΕ ε, οξύνουν και παροξύνουν την κακώς νοούμενη ε, ξενοφοβία και που δεν έχει καμία θέση εδώ και η Ευρώπη δεν θα πρέπει να δίνει τέτοια εικόνα για την υποδοχή των μεταναστών. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Ευχαριστούμε. Κυρία Σαφτιέ. Κοιτάξτε, εμείς ε, ακολουθούμε τη σειρά των συντονιστών όπως το γνωρίζετε. Αν όμως απουσιάζει ο συντονιστής, ε, τότε θα πρέπει να μας ενημερώνετε για το ποιος του αντικαθιστά. Αυτό κάνουμε συνήθως, έτσι εργαζόμαστε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και εξαιρέσεις βέβαια, αν επιμένετε. Να δώσω όμως τώρα το λόγο στον κύριο Μαν, ο οποίος είναι σκιώδης ηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή την ακρόαση σήμερα εδώ οι έξι εμπειρογνώμονες ε, κατέστησαν σαφές κυρίως το ένα, όχι τι θα πρέπει να κάνουμε, αλλά τι κάνουν οι ίδιοι στα κράτη-μέλη. Ποια είναι η πραγματικότητα σε διάφορα επίπεδα, πώς λειτουργούν οι Ο κύριος Μιούλερ ξεχάρισε πάρα πολύ ε, τι κάνει η γερμανική υπηρεσία. Είναι στρατηγική, δεν είναι ακτιβισμός. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό, ε, χρειαζόμαστε περισσότερα να κάνουμε. Χρειάζεται το χρόνο του αυτό όμως και το σύστημά του. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και από αυτά που ακούω και ε, αυτά δεν τα κάνουν μόνο οι υπάλληλοι, οι υπηρεσιακοί, αλλά πάρα πολλοί εθελοντές άμεση που ε, χωρίς τη δουλειά τους δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αυτά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προς την κυρία Ακάρη. Ε, Έχω πάει σε καταβλισμούς, έχω πάει και σε ξενώνες για συνόδευτους πρόσφυγες, έχω μιλήσει με σύρους και ε, μου λένε όταν φτάσουν και λένε ότι ε, πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα, ε, η οικογένειά μου είναι στο Χαλέπι και εγώ ένα θα ήθελα να βλέπουν οι, οι εξτρεμιστές ε, και οι ακραίοι ε, στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν με τον τρόπο αυτό τον ελεηνό τους ανθρώπους να έρθουν εκεί στους ξενώνες να δούνε. Δεν είναι εμπόρευμα αυτοί, είναι άνθρωποι. Θα ήθελα ε, να πω ότι είμαι ευγνώμων προς όλους εκείνους που φροντίζουν να γίνουν αλλαγές. Για την εκμάθηση της γλώσσας από την αρχή επιτέλους κάτι άλλαξε και το θέλουν και οι άνθρωποι. Υπάρχουν χώρες όμως που λέγουν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος οι δικαιούχοι να μην είναι ε, κάτι ε, δωρεάν. Και εκτός από την εκμάθηση της γλώσσας θα πρέπει να ξέρουν και ποιες είναι οι αξίες της κοινωνίας. Τι σημαίνει για μας η ανοχή, η ανεκτικότητα, πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία. Αυτό δεν το ξέρουν από τις δικές τους χώρες. Εμείς πόσο ε, μεγάλη σημασία δίνουμε στην αποδοχή των μειονοτήτων, για να μην πω πόσο ψηλά έχουμε το ρόλο της γυναίκας. Άρα, δεν θα πρέπει απλώς να ξέρουν μια γλώσσα και να μπορούν να ενταχθούν σε μια αγορά εργασίας για να δουλεύουν, αλλά είναι σε θέση να κατανοούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται παράλληλες κοινωνίες. Όχι στους αποκλεισμού, όχι σε ξεχωριστές ζώνες, χωριστές ζωές. Το δεύτερο θέμα που μας απασχόλησε μας ε, θα πρέπει ε, να εξαιρεθούν από τον κατώτατο μισθό. Μα τι είναι αυτό, αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός. Από μια έχουμε τους εργαζομένους ε, και από την άλλη έχουμε τους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να φέρουμε αντιπέτωπες αυτέ τις ομάδες. Θα πρέπει να πληρώνονται με τις σωστέ αμοιβέ και οι άνθρωποι αυτοί και όχι τέτοια πράγματα. Και μια ερώτηση ακόμα. Έχουμε μερικά κράτη-μέλη, το είπε και ο κύριος Μιούλερ, που θέλουν να ξέρουν ποιε είναι οι δεξιότητε και τα προσόντα του καθενό, ακόμα και αν δεν έχουν τα τυπικά προσόντα. Ότι εσεί έρχεστε εδώ, έχετε εμπειρία, έχετε γνώσει, έχετε πολλά, αλλά σε πολλέ περιπτώσει δεν αρκούν όλα αυτά που ξέρετε. Γι' αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε και θέσει μαθητεία ή άσκηση. Πολλοί νέοι με του οποίου μίλησαν μου είπαν θέλουμε γρήγορα να βρούμε δουλειά. Το κατανοώ. Και είναι και προφανέ γιατί. Γιατί θα πρέπει να στέλνουν χρήματα ε, σε εκείνους που έμειναν πίσω και τους ε, επέτρεψαν να ε, έρθουν μέχρι εδώ και μέχρι τη Γερμανία. Αλλά χωρίς εκπαίδευση και χωρίς λογική άσκηση και μαθητεία, όπου να ξέρει ο καθένας τι γίνεται και τι δεξιότητες και προσόντα έχει, δεν γίνεται δουλειά. Δεν είναι καμιά στρατηγική αυτή άμυνα ή απόκρουση ή οτιδήποτε απόρριψη για να έχουν μια πραγματική τύχη και ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Θα του το πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική δουλειά σας. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάν. Ο κύριος Μπάλα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο από τον ENF, από το ENF, τον κύριο Μαχτά, ο οποίος για παράδειγμα μας είπε ότι οι πρόσφυγες ε, σήμερα ενδεχομένω να μεσά του να έχουν και κάποιου τρομοκράτε. Ωραία, ναι, είμαστε προσεκτικοί. Και είπε επίση ότι μία απόδειξη ήταν οι τρομοκρατικέ επιθέσει του 2015 και φαντάζομαι ότι αναφερόταν στη δική μου τη χώρα, τη Γαλλία. Να του υπενθυμίσω όμω ότι αυτά τα οποία συνέβησαν στη Γαλλία το 2015 και οι δολοφόνοι που είχαμε τελικά εκεί στι τρομοκρατικέ επιθέσει δεν ήταν πρόσφυγε, ήταν ε, άνθρωποι που είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, γενικά στην Ευρώπη. Επομένως καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με πρόσφυγες και πραγματικά θέλουμε να δίνουμε μαθήματα στους συμπολίτε μας, τότε μη συγχαίουμε τα πράγματα, πράγματα εντελώς διαφορετικά. Επίσης, ο κύριος Μαχτά αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να ακούμε και τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Μα δούμε λίγο τι δημοσκοπήσει που γίνονται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι ο ίδιο ο ευρωπαϊκό λαό, οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν οριμάσει πολύ περισσότερο και είναι πιο έτοιμοι να καταβάλουν προσπάθειες από τους ίδιους τους πολιτικά ηθήνοντες, που πολλές φορές με δημογικούς τρόπους προσπαθούν να κινήσουν προς τη μία την άλλη πλευρά την ε, κοινή γνώμη. Είναι προφανώς ε, σημαντικό να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ναι, βέβαια, θέλουμε να σταθροποιήσουμε την κατάσταση στο Ιράκ και στη Συρία, αλλά καταλαβαίνετε ότι στην υφιστάμενη δύσκολη κατάσταση, στην υφιστάμενη κρίση, δεν μπορούμε ποτέ να λέμε στους ανθρώπους αυτούς ότι κοιτάξτε, ή ακόμα αν δούμε την υποσαχάρη Αφρική, δεν μπορούμε να πούμε στους πρόσφυγες αυτούς, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλώς επιστρέψτε στις χώρες σας. Υπάρχει πρόβλημα, διακόπτη πρόεδρος, πρόβλημα με τη διερμηνία. Όλες τις γλώσσες από ό,τι μου λένε. Αποκαταστάθηκε, αποκαταστάθηκε. Συνεχίστε παρακαλώ κύριε Μπαλάς. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνες οι δηλώσεις αυτές, γιατί κύριε Μαχτά, στην πράξη τι βλέπουμε. Υπάρχουν όντως κάποιες ανησυχίες, αλλά εσείς απέναντι αυτές δεν δίνετε καμία απολύτως απάντηση. Επικρίνεται και αποδοκιμάζεται απλώς κάποιες αποφάσεις χωρίς να μας λέτε τι θα πρέπει να κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική, εφόσον αναφέρεται στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Αν οι ίδιοι ευρωπαϊκοί λαοί θεωρούν ότι η κοινωνική αυτή ένταξη των προσφύγων αυτή τη στιγμή μπορεί ενδεχομένως να συνοδεύεται από αθέμητο ανταγωνισμό πιο χαμηλή μισθή για παράδειγμα για τους πρόσφυγες και ότι απειλούνται τελικά και οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες όσον αφορά το κοινωνικό τους καθεστώς και το επαγγελματικό τους καθεστώς, τότε στην περίπτωση αυτή πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί ένας απέσιος ρατσισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύει εξή αρχή, ότι η αγορά εργασίας είναι ισότιμο δικαίωμα για όλους και επομένω θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση σε ευρωπαϊκέ χώρε για το ζήτημα αυτό, προκειμένου να μπορούμε αξιοπρεπώ όλε οι χώρε να δεχόμαστε πρόσφυγε, αλλά οφείλουν και οι πρόσφυγε και εμεί να καταβάλουμε προσπάθειε για την κατάρτισή του, για την ισότιμη αναγνώριση των δεξιοτήτων τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να δεχθούμε ένα προλεταριάτο το οποίο θα πληρώνεται λιγότερο από τους Ευρωπαίους πολίτες και το οποίο θα δημιουργήσει όντως μια πολύ κρίσιμη, άσχημη κατάσταση. Το λόγο έχει η Χέλγα Στίβενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες. Πάρα πολύ ωραία τα είπατε και έχω μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το πώς μπορεί κανείς να κάνει πραγματική πολιτική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη. Και ιδιαίτερα ευτυχής με ε, αυτό που ακούσαμε για μια εγκάρσια ε, οριζόντια συγγνώμη, ε, προσέγγιση. Η ακρόαση αυτή μπορεί να είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που ακούω ότι η ένταξη είναι κάτι που συνδέεται όχι μόνο με δικαιώματα αλλά και με υποχρεώσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ένταξη των προσφύγων αλλά να περιμένουμε και από εκείνους να καταβάλουν προσπάθεια. Πρώτη ερώτηση. Πώς θεωρούν οι εμπερογνώμονες και ποιε θεωρούν ότι είναι υποχρεώσει ε, των προσφύγων και τι θα πρέπει να καταβάλουν εκείνοι ως προσπάθειες για να ενταχθούν. Επίσης μου άρεσε αυτό που άκουσα, ότι δεν υπάρχει ένας ενίο ορισμός του πρόσφυγα. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστό, έχει την ιστορία του και την πορεία του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να κοιτάμε και τα ατομικά προσόντα, τι δεξιότητε, ε, τι γίνεται και πώς αυτό ε, συνδυάζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κάτι που δεν άκουσα από τις τοποθετήσεις είναι πώς θα δοθεί ιδιαίτερη ε, μέρημνα στους ανθρώπους με αναπηρίες. Και μια δεύτερη ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε προόδου στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα σας παραπέμπω στην κατάσταση των κοφών και των κοφαλάλων ε, προσφύγων γιατί δεν ξέρουν, δεν ενημερώνονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στην ε, πληροφορία και υπάρχουν και άλλοι ανάπηροι από χώρε αφρικανικές, από χώρες ε, αραβικές που έχουν πολύ χαμηλή μόρφωση σχεδόν καθόλου λόγω των συστημάτων που επικρατούν στις χώρες αυτές και δεν είναι καθόλου εύκολο να ενταχθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κοφοί πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση σε ειδική εκπαίδευση κομμένη και εραμένη στα μέτρα τους και συγκεκριμένη κατάρτιση. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που χωλαίνει και σε πολλές χώρες και στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες. Επίσης, θα πρέπει το συντομότερο οι κοφοί πρόσφυγες να έρχονται σε επαφή με τους ε, κοφούς ε, της χώρας. Να μαθαίνουν τη νοηματική γλώσσα τη γλώσσα της χώρας για να μπορούν να εντάσσονται καλύτερα. Όπως το κάνουν και οι ε, πρόσφυγες ε, που ακούν, που μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας. Στη συνέχεια, ε, ποιες είναι οι ειδικέ προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε γενικά για ανθρώπους με αναπηρία και ιδιαίτερα τους κοφούς και κοφαλάλους. Ε, συνεργάζονται οι διάφορες οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία. Ποιες είναι οι εμπειρίες, ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές. Τι γίνεται στην Ευρώπη για να υποστηρίξουμε την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, των προσφύγων με αναπηρία. Και τέλος, θα πρέπει πολύ γρήγορα να γίνεται αυτή η δουλειά. Σήμερα είναι πάρα πολύ μακροχρόνια η διαδικασία, αλλά πρέπει να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Αυτό που ισχύει για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα σήμερα είναι αρκετά ε, βραχή διάστημα και θα πρέπει να γίνονται εντός του διαστήματος αυτού για να προχωρούν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέβενς. Ο κύριος Σούλτσε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν να μας μιλήσουν. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση. Πριν διατυπώσω την ερώτησή μου, για να μην αφήνουμε εσφαλμένες εντυπώσεις, θα ήθελα να απαντήσω σε έναν συνάδελφο. Η Γερμανία δεν χρειάζεται τους πρόσφυγες επειδή έχει δημογραφικό πρόβλημα. Η Γερμανία χρόνια πριν ξεκίνησε μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Κοιτάξτε λίγο την Agenda ε, 2010 με τον Gerhard Σρόντερ τότε ως καγκελάριο. Θα μάθετε πολλά πράγματα και μπορεί και να ξανασκεφτείτε ορισμένε θέσει σας. Δύο πράγματα λοιπόν. Ελάχιστος μισθός καταρχάς και συνέπεια στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα θα απευθύνω την ερώτηση στον κύριο από τη Γερμανία. Εγώ δεν υποστηρίζω την ιδέα της ε, αυτόματης ε, κατάργησης για τον εργαζόμενο πρόσφυγα ή μετανάστη του ελάχιστου μισθού. Από την άλλη, στη δική μου την περιοχή έχουμε 10% ε, ανεργία, περισσότερο βέβαια από το μέσο όρο της Γερμανίας. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα ήθελαν να αναλάβουν δράση και να προσλάβουν και πρόσφυγες, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να καταβάλουν τον ελάχιστο μισθό στους μετανάστες ή πρόσφυγες, γιατί αυτοί δεν έχουν πάντα τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και μήπως τελικά μέσα από το θέμα αυτό του ελάχιστου μισθού ε, μπορέσουμε, εάν αρθεί δηλαδή η προσφυγε γιατι αυτοι δεν εχουν παντα τις απαιτούμενε δεξιοτητες και γνωσεις ειναι κατι λοιπον το οποιο πρεπει να συζητηθει και μήπω τελικα μεσα απο το θεμα αυτο του ελάχιστου μισθού, θα μπορούσαμε να ε, καταπολεμήσουμε την παράνομη εργασία και να επιτρέψουμε σε ανθρώπους που έχουν πολύ πολύ περιορισμένες δεξιότητες ή δυνατότητες απασχόλησης να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ δύσκολο να σωματωθεί κανείς ε, στην αγορά εργασίας στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν ίσως θα ήταν μια αναστολή του ελάχιστου μισθού, όπως ισχύει στη Γερμανία για τους μακροχρόνια ανέργους, ε, να βοηθήσει στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και βέβαια να διευκολύνει και σε γραφειοκρατικό επίπεδο και επίσης σε σχέση με την επαλήθευση όταν πρόκειται δηλαδή για τη δυνατότητα απασχόληση ενός πρόσφυγα, την υποχρέωση για την ε, ε, υπηρεσία να επαληθεύσει ότι δεν θα μπορούσε αντίστοιχα να έχει απασχοληθεί ένας ε, εγχώριος άνεργος. Θέλετε να μας πείτε κάποιες ιδέες και αν αυτό μπορεί να βοηθήσει, αν μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, ε, να βοηθήσει και βέβαια και τον πρόσφυγα στην ενσωματωσή του. Και κάτι ακόμη, το οποίο μας απασχολεί στη Γερμανία και πρέπει να συζητηθεί γενικότερα, ε, η κοινωνική χρηματοδότηση ή γενικότερα τα κονδύλα τα οποία έχουμε από την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επί παραδείγματι, η κυρία Τάισεν, η Επίτροπος, πρόσφατα σε μια συνεδρίαση ερωτήθηκε για το πώς μπορούν τα κοινωνικά κονδύλια να αξιοποιηθούν για την ενσωμάτωση και την, κοινωνική, και την επασχόληση των μεταναστών. Ε, μας είπε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ότι μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί. Ερωτώ λοιπόν εσείς αυτά τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά, του Κοινωνικού Ταμείου και αντίστοιχα, πώς τα αξιοποιείτε και νομίζετε ότι θα μπορούσατε να έχετε κάποια καλύτερη ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάσλιβιέκα για αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, στους προσκεκλημένους μας γιατί έφτασα με καθυστέρηση στη συνεδρία αλλά είχαμε ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή όπου έπρεπε να είμαι παρούσα. Ζητώ συγγνώμη γιατί γνωρίζω ότι το θέμα των προσφύγων είναι άκρο σημαντικό και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Και διαπιστώνω πως καμία πλευρά δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στις διαστάσεις που εκδηλώνεται στην Ήπειρό μας. Η Ελίζα υπεγράμμισε κάτι πολύ σημαντικό. Πώς οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι καταρτίζουν, ενημερώνουν τους πρόσφυγες, πώς μπορεί αυτοί να στηριχθούν. Και ιδιαίτερα διαπίστωσα το καλοκαίρι όταν έφταναν στην Ουγγαρία οι πρόσφυγες και τους εγκαθιστούσαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ε, αισθάνονταν δυσφορία γιατί οι ότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στην Ευρώπη. Δηλαδή έλεγαν ότι θα έρθουμε στην Ευρώπη πρέπει να μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό νομίζω αποτελεί μία ένδειξη ότι οι υπηρεσίες που είχαν να διαχειριστούν τους ε, αφυγνούμενους πρόσφυγες δεν ήταν έτοιμες να τους εξηγήσουν ότι υποβάλλουν αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα και ότι βρίσκονταν μέχρι την υποβολή της σχετικής αιτήσεως παράνομα σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Ερωτώ λοιπόν, εσείς κάνετε κάτι για να ενημερώσετε τους πρόσφυγες. Δεν πρέπει να του ενημερώνετε από την πρώτη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι του Ευρωπαϊκή Επικράτεια ή οποιοδήποτε άλλο κράτο. Δεν πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά του, αλλά και για τι υποχρεώσει του, για το πώ θα πρέπει να προετοιμάζονται. Η απουσία τέτοια ενημέρωση, πιστεύω, προξενεί αισθήματα δυσφορία και δυσκολεύει και την, αντι... την αντίληψη από πλευρά των προσφύγων της κατάστασης. Τους κάνει να ζητούν πράγματα στα οποία δεν έχουν δικαίωμα. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και ενίσχυση των εντάσσεων και της επιθετικότητας από τις δύο πλευρές. Ενώ θα έπρεπε να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε ένα τον άλλον. Εξού και η δεύτερη ερώτηση. Η ευρωπαϊκή κοινωνία πώς μπορεί να προετοιμαστεί ώστε να αντιληφθεί αλλά και να δεχθεί την κατάσταση. Εγώ προερχόμαι από την Πολωνία χώρα η οποία δεν έχει καμία εμπειρία όπως αντίστοιχα η Γαλλία και η Ιταλία από υποδοχή προσφύγων και ιδίως προσφύγων από την Αφρική. Οι καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίσαμε στο Παρίσι και την Κολονία δείχνει ότι οι πολίτες φοβούνται. Φοβούνται. Και οι τοπικές κυβερνήσεις, σχολεία κτλ. δεν είναι καν έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτές τις αφήξεις γιατί θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε στους κατοίκους, να τους βοηθήσουμε, να τους πείσουμε οι δυνατόν ότι υπάρχει ότι είναι σκόπιμο να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε όλοι μαζί. Ελπίζω να το προσέχετε και σε αυτό, στα διάσταση, σε μια χώρα όπως η δική μου που δεν έχουμε καμία ανεμπειρία από την ενσωμάτωση ξένων. Γιατί η ενσωμάτωση θα έπρεπε να ε, είναι κάτι το οποίο επιδιώκουν και οι δύο πλευρές. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε. Ο κύριος Χοκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ είμαι Πολωνός. Αλλά έχω διαφορετικές θέσεις. Ε, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα και απαραίτητη αυτή η συζήτηση, ωστόσο δεν με καθησύχασε η ακρόαση που κάναμε. Του αντίον βλέπω μόνο ευσεβείς πόθη να εκφράζονται, ενώ όλα αυτά φαίνονται πολύ ωραία, η ενσωμάτωση, η υποδοχή, η παροχή υποστήριξης. Μπορεί να φαίνονται πολύ ωραία, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και πολλές φορές πολύ τραγική και για τον ε, πρόσφυγα και για τον κάτοικο της Ένωσης. Η κάθε χώρα έχει τη δική της εμπειρία, την ιστορία της, την εθνική της ταυτότητα. Ενσωμάτωση χωρίς ε, ε, αφομοίωση είναι ουτοπία και το επαναλαμβάνω, είναι συνιστά ουτοπία. Θα ήθελα να επενθυμίσω την, το τάγμα της, του ελέους Orden Caritatis που σημαίνει πρώτα προσφέρουμε αγάπη και ασφάλεια στην οικογένεια, στη συνέχεια στη βατρίδα και μετά στις άλλες κοινότητες. Και επίσης πώς θα γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ του καθεστώτος του πρόσφυγα, του μετανάστη, του ετούντος στο άσυλο, πού θα σημειωθούν τα όρια. Κοιτάμε παραδείγματι τους λόγους της μετανάστευσης. και πόσα εκατομμύρια μετανάστες πρέπει να φτάσουν να μεταναστεύσουν μέχρι ότου τεθεί ένα τέρμα στη μετανάστευση. Επίσης η κατάσταση στην αγορά εργασίας πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε φανταστές λύσεις για τα προβλήματα που έχουν οι δικές μας χώρες. Και για να ολοκληρώσω, ναι, είναι απαραίτητο να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά, αλλά πολύ πιο απαραίτητο είναι να αναλάβουμε συγκεκριμένε δράσει και ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμούμαστε ότι οφείλουμε να προσφέρουμε βοήθεια στους ανθρώπους στην πηγή του προβλήματο. Πρέπει να μα απασχολήσει η αντιμετώπιση της ρίζας, της αιτίας και όχι του αιτιατού. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για μα. Ποτέ δεν θα υπάρξει πλήρης αφομοίωση ή ενσωμάτωση εάν δεν ελαχιστοποιήσουμε τους ίδιους τους λόγους της μετανάστευσης. Ευχαριστώ Μάγερ. Ατζέα. Ατζέα παρακαλώ. Πραγματικά κυρία Πρόεδρε είναι πολύ δύσκολο να πάρω το λόγο τώρα μετά από όλα αυτά τα οποία άκουσα. Ειλικρινά Ποιος ο λόγος να είναι κανείς βουλευτής, ευρωβουλευτής σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί 28 κράτη-μέλη εντελώ διαφορετικά μεταξύ τους, μιλώντας κατά της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δούμε λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας. Να αφήσουμε τη δική μας την ησυχία και βλέπω ότι κάθε φορά που το κάνουμε αυτό το πράγμα πανικοβαλόμαστε τελικά. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για διαφορετικές μορφές συμπάθειας ή αγάπης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για διαφορετικές μορφές αγάπης. Η αγάπη είναι μία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή μέσω της ενσωμάτωσης, μιλώντας για ενσωμάτωση, να αφήνουμε εκτός κάποιους ανθρώπους. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε δεν υπάρχει καν λόγος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί το μοντέλο της ενσωμάτωσης και της ένταξης ενδεχομένως επειδή είμαστε εντελώς κλειστοί και ανίκανοι τελικά να δούμε πέρα από τη δική μας τη μύτη, πέρα από τη δική μας τη χώρα. Είμαστε σαφώς 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προτάθηκε στην Βαλέτα μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση και για την ενσωμάτωση των προσφύγων, Τότε ήμασταν όλοι εκεί, πολύ ωραία, αξιοπρεπείς και με ιδιαίτερη χαρά είπαμε ναι, ναι βέβαια, να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή, να ελοποστηριχθούμε, να τους υποδεχθούμε τους πρόσφυγες αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία εβδομάδα αργότερα άρχιζε κάθε χώρα ξεχωριστά να χτίζει το δικό της το τείχος. Επομένως η αρχή αυτή της αλληλεγγύης στην πράξη δεν εφαρμοζόταν. Πολύ ωραία λοιπόν. Πολύ καλοί είμαστε στα λόγια. Όταν χρειάζεται όμως τα λόγια να τα κάνουμε πράξη, τότε πραγματικά μένουμε τραγικά στάσιμοι. Δεν έχουμε δει πιο τραγική στασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα αυτό κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται ένα μη πρόβλημα θα μπορούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα τόσα εκατομμύρια κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούμε να σωματώσουμε το μεγάλο αυτό αριθμό των προσφύγων. Αλλά αν αυτή τη στιγμή αφήνεται ορισμένε μόνο χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση, προφανώ δεν μπορούν να τα καταφέρουν και προφανώ δεν μπορούμε να έχουμε ένταξη και ενσωμάτωση. Και προφανώ γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες στους ανθρώπους αυτούς, ισότιμες με τις συνθήκες που έχουμε για τους υπόλοιπους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού πάνε οι άνθρωποι αυτοί, πόσοι έχουν τα κέντρα υποδοχής, ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσής τους. Ας τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα, από πού φτάνουν καταρχάς οι άνθρωποι αυτοί. Και ας κάνουμε και μία διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν πόλεμο και στους τρομοκράτες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερη σύγχυση από το πράγμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αποφύγουμε τη σύγχυση αυτή και να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πιο μακριά από τη δική μας τη μύτη και από τη δική μας τη χώρα. Βλέπω εγώ την κατάσταση στην Ιταλία, μια χώρα που έζησε αντίστροφα την κατάσταση. Στο Βέλγιο Υπάρχει μια πολύ μεγάλη Ιταλική κοινότητα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη βελγική κοινωνία και θεωρώ ότι έχουμε επιφέρει, έχουμε προσθέσει μια προστιθέμενη αξία όταν ήρθαμε ως Αθρακορίχη στο Βέλγιο. Αλλά ακόμα και στην Πολωνία δούμε τα πράγματα. Οι Πολωνοί μετανάστες μια χαρά ενσωματώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Επομένως δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να λέτε τι σημαίνει ενσωμάτωση, τι σημαίνει ένταξη, γιατί οι ίδιοι τη ζήσατε. Οι ίδιοι παππούδες σας, όπως οι δικοί μου παππούδες, βίωσαν την κατάσταση αυτή. Προφανώς όταν φύγαμε από την ε, Ιταλία και πήγαμε σε άλλες χώρες δεν μας αντιμετώπισαν πάντα θετικά, αλλά αποτελέσαμε τελικά μία πηγή και με τον ένα τον άλλο τρόπο, μία προστιθέμενη αξία, με τον ένα τον άλλο τρόπο τελικά ενσωματωθήκαμε. Νομίζω λοιπόν ότι Πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε, εμπνεόμενοι από τα παραδείγματα αυτά του παρελθόντο, πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορούμε όμω να θελοτυφλούμε λόγω του φόβου αυτή τη στιγμή και δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε απλώ εδώ πέρα και να, να σε θεωρητικέ κουβέντε. Η κυρία Κιέγγε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την πολύ σημαντική αυτή συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα και μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε περισσότερο, να κάνουμε αντιπαράθεση απόψεων και να δούμε τελικά τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Λυπάμαι που έφτασα καθυστερημένη, είχαν λυμμένε υποχρεώσει και σε άλλε επιτροπέ. Παρ' όλα αυτά θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρω να παραστώ έστω και καθυστερημένα στην ακρόαση αυτή. Και νομίζω ότι πραγματικά οι παρουσιάσει ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Εγώ είμαι συγγήτρια έκθεσης πρωτοβουλίας για μια ολιστική προσέγγιση του φαινομένου της μετανάστευσης στη Μεσόγειο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα γιατί το ζήτημα της μετανάστευσης και το ζήτημα της ενσωμάτωσης αντιμετωπίζεται και στη δική μου την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα τις μεταναστευτικές ροές, το μεταναστευτικό φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν προωθήσει την κινητικότητα ταλέντων, γνώσης και ανθρώπων θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις πάρα πολλές ε, που καλείται αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσει λόγω τη δημογραφική εξέλιξη τη και λόγω των πολύ μεγάλων κενών που υπάρχουν πολύ συχνά στην αγορά εργασία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένου κοινού κανόνε για την νόμιμη είσοδο των μεταναστών από τι τρίτε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα όσον αφορά την οικονομική μετανάστευση, είμαστε κατά οποιασδήποτε επαγγελματικής εκμετάλλευσης των μεταναστών και των προσφύγων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπονται κυρώσει. Μόνο το φαινόμενο αυτό τελικά συνδέεται με φαινόμενο εμπορία ανθρώπων. Θέλουμε εμεί ε, η ε, οδηγία 52 κάθος 2009 τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, να προστατεύει επίσης και τα θύματα της ε, εμπορίας ανθρώπων που πέφτουν στη συνέχεια θύματα επαγγελματικής εκμετάλλευσης. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό θα κάνει και μία πρόταση. Συμμετέχω επίσης και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε και μία ακόμα πρόταση, την μπλε κάρτα. Χρειαζόμαστε εδώ πέρα μία πιο φιλόδοξη πρόταση για την ενσωμάτωση των εργαζομένων, των προσφύγων με συγχωρείτε στην αγορά εργασίας. Το να καταφέρουμε να έχουμε νόμιμες οδούς για τους μετανάστες στην ευρωπαϊκή επικράτεια θα πρέπει να συνοδεύεται από έντονα πολιτικά μέτρα τα οποία έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση των μεταναστών και να προβλέπεται στη συνέχεια και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσφύγων και των μεταναστών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μέσω της ενσωμάτωσης και της έντοξης μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο σημαντική μας πρόκληση λοιπόν, κοινή πρόκληση αυτή τη στιγμή, είναι να έχουμε μια προσέγγιση στη μετανάστευση που θα έχει ως βασική προτεραιότητα την ενσωμάτωση των προσφύγων στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ισχύουν και για αυτούς ανάλογες συνθήκες με αυτές που ισχύουν και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικότερο εργαλείο της ενσωμάτωσης είναι η απασχόληση, είναι η δουλειά, η εργασία. Και γι' αυτό το λόγο ζητούμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά το άρθρο 15 της Οδηγίας για την Υποδοχή και κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουν ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αναφέρομαι εδώ πέρα σε πρόσβαση. Μετά από εννιά μήνες αφότου υποβάλλουν την αίτησή τους. Αναλύσαμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και άκουσα και κάποιες παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν στο πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Αναλύσαμε λοιπόν το σύστημα του ασύλου, βλέποντας πραγματικά πώς έχουν τα πράγματα και θελώντας τελικά εδώ πέρα να δούμε ποιο θα είναι το αρμόδιο κράτος μέλος, το οποίο θα πρέπει να ασχολείται με το ζήτημα των οικογενειακών δεσμών και επομένω της οικογενειακής επανένωσης. Και δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο στην πράξη. Δεν εντοπίζεται δηλαδή το σωστό κράτο μέλο το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί με την οικογενειακή επανένωση, γιατί ακόμα ισχύει ο κανόνα τη χώρα, τη πρώτη χώρα πρόσβαση, ένταξη. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και την ρήτρα της διακριτικής μεταχείρισης. Τα ζητήματα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Οφείλουμε να εμβαθύνουμε επίσης την κατάσταση των μεθοριακών κρατών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση εξαιτίας επειδή θέτουμε ένα αμφιβόλο την ελεύθερη κυκλοφορία των μεταναστών στο χώρο Σέγγεν. Αυτό θα έχει πολύ δεινέ συνέπειε όχι μόνο για του μετανάστε, αλλά και για του ίδιου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στου ίδιου εργαζόμενου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επηρεάσει τελικά την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, αλλά και την ελεύθερη κυκλοφορία των ίδιων των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει πολύ σοβαρά να στοχαστούμε όλα αυτά τα ζητήματα και να καταφέρουμε να ενημερώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ίδιου του πολίτες μας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ του ομιλητέ όλου για τι ερωτήσει και τι παρεμβάσει του. και δίνω το λόγο τώρα στους προσκεκλημένους μας. Πάρα πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα ή εάν... Έχετε κάτι πιο καινούριο να απαντήσετε. Πρώτα, η κυρία που εκπροσωπεί τους Σύρους πρόσφυγες, και την πρωτοβουλία Μαρίνστατ. Ναι, βεβαίως. Απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε ερωτήσει. Και να δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα για τους Ευρωπαίους που δεν έχουν δουλειά. Και μιλάμε για ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των προσφύγων. Ίσως αυτό ακούγεται για ορισμένου ότι θέλουμε να δώσουμε την προτεραιότητα στου πρόσφυγε. Θα απαντήσω το εξή λοιπόν εδώ, το να δώσουμε σε πρόσφυγε τα εργαλεία να εγκαταστούν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασία σε σχέση με άλλου. και μετά να αντιμετωπίσουμε το, να αντιμετωπιστεί μάλλον το όλο πρόβλημα της ενεργείας ε, σαν σύνολο είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπουν στην αγορά εργασίας γιατί θέλουν να κερδίσουν χρήματα όχι μόνο για να πληρώσουν αυτούς που τους βοηθούν να έρθουν στην Ευρώπη, αλλά και για να μετατραπούν σε ε, νομοταγείς φορολογούμενους, να, κάνουν, ε, να συμβάλλουν στις οικονομίες των χωρών που τους υποδέχονται με ίσους όρους και όχι απλώς να είναι αποδέκτες επιδοτήσεων. Να ρωτήσετε έναν πρόσφυγα σε ένα καταβλισμό τι χρειάζεται, θα σας απαντήσει τρία πράγματα χρειάζομαι. Γλώσσα, ενημέρωση τι συμβαίνει στη χώρα ή τι θα συμβεί στο μέλλον, στη χώρα μου, θα συμβεί στο μέλλον και η αδίποτε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ακόμη και με εθελοντική εργασία. Ο ετών το άσυλο στην Σουηδία έχει την άδεια να εργαστεί. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ακόμα και όταν έχουν τη δυνατότητα της εργασίας οι πρόσφυγες, οι επίπτες άσυλο, δεν τους δίνουν δουλειά γιατί υπάρχουν άλλες ανησυχίες και μιλήματα. Και επίσης δεν θέλω ε, να ε, παρουσιάσω την κατάσταση να είναι σε αντιπαράθεση ο πρόσφυγας με τον με τον άνεργο που είναι στη θέση εργασία. Πολλές φορές όμως ο εργοδότης δεν δίνει δουλειά στον... δεν, δεν ανοίγει μια θέση εργασία, γιατί του κοστίζει πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και ίσως θα ήταν καλό να βρούμε ένα σχέδιο ε, απασχόληση, εγκατάστασης στα σχολεία, στα εργαστήρια, στον τόπο στον οποίο γίνεται η βασική κατάρτιση. Δεν θα κοστίσει πιο πολύ, απλώς θα έχει μια πρακτική ε, εφαρμογή η κατάρτιση που θα προσφέρεται για το ότι θα πρέπει να επανέρχονται στις χώρες τους και να ζουν ευτυχείς οι πρόσφυγες. Έχω να δώσω δύο απαντήσεις. Πρώτον, ελπίζουμε η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της στο πολιτικό ζήτημα και να βρεθούν οι λύσεις στο Συριακό και σας διαβεβαιώ ότι πολλοί θα σταματήσουν να έρχονται στην Ευρώπη. Άπαξ και επιληθεί το Συριακό. Όσο δεν αφορά αυτούς που θέλετε εσείς να επαναπατρίσετε, παρακαλώ αποφασίστε. Τι θέλετε. Θέλετε να τους ενσωματώσετε στις κοινωνίες, θέλετε να τους στείλετε πίσω. Μέχρι να μάθετε τι θέλετε, μέχρι να αποφασίσετε τι θέλετε. Γιατί πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η πολιτική βούληση για να είμαστε απολύτω σαφέ. Και βεβαίως πολλοί θα επιστρέψουν στις χώρε του, αλλά δεν μπορείτε να υποχρεώσετε κανέναν Εάν επιλέξει κάποιος να μείνει εδώ, να ζήσει εδώ, να είναι μέλος της κοινωνίας, έτσι πρέπει να γίνει. Κάποιος που δεν μπορεί να μπει μέσα στις κοινωνίες, ας γυρίσει πίσω. Αλλά πρέπει αυτό να γίνεται θελοντικά. Και βέβαια για να μιλήσουμε για την υποδοχή και την αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, οι αντιδράσεις των τοπικών ε, φορέων όταν έρχονται και μας βοηθούν και μας υποδέχονται, κάνει και άλλους να αντιληφθούν ότι μπορεί να είναι ε, καλό αυτό. Ας το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα. Εγώ είμαι αρμόδια για ένα εγχείρημα στην περιοχή μου με τέσσερις δασκάλους, επαγγελματίες δασκάλους γλώσσας, που προσφέρουν μαθήματα 8 ώρες την εβδομάδα σε 100 σπουδαστές στα μαθήματά τους. Έχουμε ήδη φτάσει, έχουν ήδη αυτοί οι σπουδαστές φτάσει σε επίπεδο να μπορούν να εκφράζονται στην γλώσσα της ε, χώρας και να είναι έτοιμοι πάρα πολύ σύντομα να μπουν ε, επίσης ώρες στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, πολλές προσπάθειες γίνονται και χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη. Εάν οι κυβερνήσεις λοιπόν υιοθετήσουν αυτή την κοινωνική προσέγγιση και προσφορά, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Μίλες από τη Γερμανία. Federal Employment Agency, Germany, please. Three minutes. Για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις. Μια σειρά ολόκληρη. Θα κάνω ό,τι μπορώ αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ είμαι στις Βρυξέλλες. Δηλαδή είμαι στις Βρυξέλλες και ε, είμαι στη διάθεσή σας και μετά τη συνεδρίαση. Ε, πολύ σημαντικό μήνυμα και εδώ απαντώ σε πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα είναι η ίση μεταχείριση. Αυτή είναι η βάση. Δεν είναι μόνο ένα θέμα που επιβάλλει ο νόμος, αλλά έχει και νόημα από πλευράς πολιτικής ένταξη. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε απλούστατα, είτε πρόκειται για επιδοτούμενε θέσεις εργασίας, είτε πρόκειται για αναπηρικά επιδόματα, είτε πρόκειται για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσιο, είτε για κάποιε εξετάσει. Ε, σε περίπτωση που δεν αποφασίσει διαφορετικά ο νομοθέτης δεν γίνεται καμία διάκριση. Δηλαδή, αν κάποιος ε, πληρεί τα προσόντα να πάρει επιδοτούμενη θέση εργασίας δεν έχει καμία σημασία αν είναι πρόσφυγας, αν είναι Ισπανός μακροχρόνιος άνεργος ή Γερμανός μακροχρόνιος άνεργος. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Εάν πληρούνται οι προποθέσει και τα κριτήρια, τότε εμεί παρέχουμε αυτή την υπηρεσία εγγυημένη. Το ίδιο ισχύει και με τι εξαιρέσει για το κατώτατο ημερομίσιο αλλά όλα αυτά τα πράγματα τα έχει ορίσει ο νομοθετής και μας δίνει το περιθώριο ε, στο οποίο εμείς κινούμαστε και εκτελούμε. Και την αναπηρία τη χρησιμοποιώ και τη δανείζομαι ως παράδειγμα γιατί έχουμε ειδικέ ομάδες που ασχολούνται με άνθρωπους με αναπηρία και όχι μόνο αναπηρία, έτσι και, ψυχική και διανοητική ε, αναπηρία με τα τραυματικά σοκ και τα λοιπά. Αυτά υπάρχουν ήδη στην κοινωνία, δεν τα φτιάξαμε τώρα που ήρθαν οι πρόσφυγες. Ε, ε επίσης, η υποχρέωση... Ε, στέγης και παραμονής υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Υπάρχει κίνδυνος γετοποίησης και δεν μιλώ εδώ γενικά για τις αστικές περιοχές. Ακούσαμε για τις πολυκατοικίες και τα μεγάλα συγκροτήματα στα προάστια ε, των γαλλικών πόλεων αλλά το θέμα είναι τι δραστηριότητες ασκεί κανείς, ποιο είναι το περιβάλλον και τι μισθό παίρνει. Τα προσωπικά δίκτυα Βέβαια, κάθε ένταξη στην εργασία, ιδιαίτερα για τους μετανάστες, είναι ένα θέμα που αναλαμβάνουν τα δίκτυα. Οι βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν και γίνονται και ανταλλαγές διμερείς όμως με τον εκάστοτε ΟΑΕΔ, ας πούμε, της κάθε χώρας. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, υπάρχει θεσμική συνεργασία και ε, η δική σας απόφαση για να συσταθεί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά έχουμε επίσημη ε, ανταλλαγή απόψεων και ομάδα εργασίας και μας απασχολεί τακτικά στις συνεδριάσεις μας. Καταγραφή των προσόντων και των δεξιοτήτων. Τρία πράγματα, οπτικά είναι αυτά. Έχουν να κάνουν πάρα πολλά με εικόνες, πρακτικά και με φωτογραφίες στην αγορά εργασίας και στον τόπο δουλειάς και online. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω να σας τα πω για λόγους χρόνου. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος ε, Αβώ από τον Ερυθρό Σταυρό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιέζει όντω ο χρόνο. Θα απαντήσω μόνο σε δύο ερωτήσει που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικέ. Όσον αφορά την έκθεση αυτή τη κυρία Στάινμπρουκ, λοιπόν, την ερώτηση, όσον αφορά την ανταλλαγή των πρακτικών και μία ακόμα ερώτηση που ακούσαμε όσον αφορά τα πρότυπα παροχή υπηρεσιών. Όντω υπάρχει μία ανταλλαγή των πρακτικών στα πλαίσια των φορέων παροχής υπηρεσιών, ευτυχώς μάλιστα, αν δει κανεί την κλίμακα τη ε, κρίση, όντω απαιτούνται αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικέ υποδομέ προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Υπάρχουν όμω δύο βασικοί περιορισμοί και θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτού. Ήδη στην παρουσίασή μου είχα πει ότι οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού παρέχουν υπηρεσίε κατά 50% στου πρόσφυγε. Το υπόλοιπο 50% παρέχεται από άλλου φορεί, όπω η Κάριτα για παράδειγμα, ή από τα ίδια τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια θα πρέπει βέβαια να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα, δηλαδή κατάλογοι συγκεκριμένων υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχονται προς τους ε, μετανάστες. Αυτό ισχύει και για τον ανθρωπιστικό τομέα, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη ένταξή του στην κοινωνία που μας απασχόλησε σήμερα. Στο πλαίσιο βέβαια του Ερυθρού Σταυρού εδώ και 150 χρόνια σε ορισμένες χώρες έχουμε ήδη ένα κατάλογο ελάχιστων υπηρεσιών που θα πρέπει να παράσχονται σε χώρες διέλευσης όπως η Αυστρία για παράδειγμα. Οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε Basic Primary Health Care, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και κάποιες άλλες βασικές υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη ούτε στο πλαίσιο των ίδιων των γραφείων του Ερυθρού Σταυρού στα εκάστοτε κράτη-μέλη της Ένωσης. Όπω είπε λοιπόν και ο κύριος Μιούλερ, εγώ βρίσκομαι στις Βρυξέλλες και είμαι προφανώς και εγώ στη θέση σας για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Thank Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Σομαχώρο. Παρακαλώ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έλεγα και προηγουμένως στην ε, παρουσίασή μου, όταν σας παρουσίασα τις τρεις διαστάσεις και τις τρεις προσεγγίσεις, πρέπει να πω ότι είναι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των βουλευτών. Αλλά αν δεν έχεις μια ελάχιστη βάση για το πώς θα προσεγγίσεις αυτά τα θέματα, είναι πολύ δύσκολο να προτείνεις λύσεις. Μέχρι σήμερα, τι έχουμε μια διαστροτική προσέγγιση. Όλα αυτά που γίνονται είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία στην οποία ζούμε. Δεν μιλώ για την Ευρωζώνη τώρα, μιλώ για τον κόσμο ολόκληρο που ζούμε, την κοινωνία μας. Που ε, ε διασυνδέονται όλες αυτές οι διαστάσεις. Άρα, το πρώτο είναι να κατανοήσουμε τι γίνεται. Το δεύτερο είναι ότι η αντίληψη που έχουμε, πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. δημιουργεί την εντύπωση ότι μας κατακλείζουν οι πρόσφυγες. Είναι 60 εκατομμύρια παγκοσμίω οι πρόσφυγες. Είναι άνθρωποι που αναγκάστηκαν για λόγους που συνδέονται με τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως, οικονομικούς ή άλλους πολέμου, που έχουν φύγει. Οι 9 στους 10 από αυτούς τους πρόσφυγες δεν ζουν στην Ευρώπη, είναι αλλού. Το τρίτο στοιχείο αφορά ε, την αγορά εργασίας. Τι μας λένε σήμερα οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και το είπα προηγουμένως, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία ε, του 2013 στο άρθρο 15 ζητεί από τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν στους πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αλλά αυτή, αυτό είναι σε εθελουσία βάση. Δεν υπάρχει τίποτα υποχρεωτικό, ούτε εναρμόνιση, ούτε δέσμευση, ούτε ελάχιστο επίπεδο για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση. Και όταν 28 οι διαφορετικές νομικές, οικονομικές, πολιτιστικές πραγματικότητες, ε, είναι προφανές ότι κινδυνεύουμε εκεί να βρεθούμε σε μία ζούγκλα. Δηλαδή, να υπάρχει ένας κατώτατος μισθός για να μπαίνουν στην αγορά εργασίας οι πρόσφυγες και εδώ υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός μεταξύ προσφύγων μακροχρονίων ανέργων και όλων των υπολείπων. Και θα πρέπει αυτό να αποφευθεί. Τελευταίο στοιχείο, βέλτιστες πρακτικές. Στην Ιταλία, εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα, Ένωση, κάναμε ένα δίκτυο γραφείων και οι φωτογραφίες αυτές που είδατε είναι στα χωράφια που εργάζονται ως, αγροτικοί, ε, ως, εργάτες γης όχι μόνο οι πρόσφυγες και ο ντόπιο πληθυσμό και ζει έτσι. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για τους πρόσφυγες, θέλουμε βελτίωση και δεν υπάρχει διάκριση πρόσφυγες και μετανάστες. πρέπει να καταλάβουμε το φαινόμενο στους ε, πραγματικού όρου. Ευχαριστώ η κυρία Βεράστ από τη Φλάνδρα. Um, first of all... Ναι, καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή. Υπόθηκε ότι δίνεται η εντύπωση που προσπαθούμε να απλουστεύσουμε την πρόκληση, να, απλο... να υποβαθμίσουμε την πρόκληση. Όχι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και το ξέρουμε πολύ καλά. 70% των προσφύγων που έχουν φτάσει στη Φλάνδρα ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να διαβάσουν καν το λατινικό αλφάβητο ή να το γράψουν. Από την άλλη όμως ξέρουμε και πολύ καλά το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι πεστροί πρόσφυγες έχουν έρθει και θα, μον... θα μείνουν μόνιμα και άρα πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα κοινό μέλλον για τους πρόσφυγες. Απασχόληση, η απασχόληση είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, ε, επιστρέψουν τη δωρεά της κοινωνίας και ό,τι τους έχει προσφέρει την προσφορά της κοινωνίας. Επίσης, οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα το οποίο οργανώνουμε εμείς Έχουμε, ε, κάνουμε με συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση, ταυτόχρονα όμως ήδη οι κανόνες ισχύουν για τους πάντες και όπως ανέφερε άλλωστε και ο κύριος Μπούχφαλτ η ενσωμάτωση απαιτεί προσωποποιημένη προσέγγιση και αυτό ισχύει οπωσδήποτε και ακόμη περισσότερο για τους πρόσφυγες με αναπηρία. Με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις λοιπόν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες με αναπηρία ώστε να παρακολουθήσουν καλύτερα το πρόγραμμα αν και πρέπει να ομολογήσω ότι οπωσδήποτε υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και εν τέλει θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχει ανάγκη να στηριχθούν και οι επαγγελματίες που εργάζονται στους πρόσφυγες. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να προσφέρουμε και συμβουλές σε επαγγελματίες από άλλους χώρους που έχουν να κάνουν με πρόσφυγες. Και βέβαια να προσφέρουμε την υποστήριξή μας και ε, την αρρωγή μας στους πρόσφυγες. Πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα παράλληλα. Ευχαριστώ Χολεβίνσκι, ειδικό τη μεταναστευτική πολιτική του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια κύρια ζητήματα ε, και παρατηρήσεις που θα ήθελα να δώσω απαντήσεις. Και καταρχά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα στην τοποθέτησή μου, ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα στους τομείς ε, στους οποίους υπάρχει μεγάλη πυκνότητα στις περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται μεγάλη πυκνότητα ε, προσφύγων και για την Ευρώπη αυτό σημαίνει και την ε, εστίαση, την παροχή μάλλον υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά εάν και το κόστος μπορεί να είναι υψηλό, αν όμως ε, τα μέτρα ενσωμάτωσης και βέβαια η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ε, προχωρήσουν ε, ταχύτατα, τότε μπορεί να περιοριστεί το κόστος. Κάθε τι βέβαια ε, κοστίζει σε χρήμα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τις γειτονικέ χώρες, εκείνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής των προσφύγων, τη μεγάλη διάσκεψη για τις Συριές, την οποία δόθηκαν υποσχέσεις από τα κράτη για 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε χορηγία, ε, όλα πρέπει να γίνουν και ταυτόχρονα και στην ισότιμη μεταχείριση. Το Διεθνέ Γραφείο Εργασία, η διεθνή Οργάνωση εργασία θέλει να υπογραμμίσει αυτήν την ε, διάσταση. Βλέπουμε σε σχέση με τους μετανάστες ε, σε ορισμένες χώρες να μην προσφέρεται ο ελάχιστος μισθός στους μετανάστες όταν προβλέπεται για τους εγχώρους εργαζόμενους. Αυτό βεβαίως ένα τα ισότιμης μεταχείρισης, αλλά ταυτόχρονα και όπως είπα και στην τοποθέτησή μου νωρίτερα, υπονομεύει τα δικαιώματα, τους μισθούς και τις συνθήκες απασχόλησης για τον κάθε ένα μέσα στη χώρα εν τέλει. Όταν λοιπόν εξετάζουμε διάφορες λύσεις για τους ε, ασκούμενους ή καταρτιζόμενους, δεν πρέπει να μετατρέπονται αυτόματα αυτοί οι ασκούμενοι σε εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά με, τον άλλο εργαζόμενο, με έναν άλλον εργαζόμενο αλλά παίρνουν λιγότερα λεφτά. Επίσης κάποιες προσπάθειες για παρεμπόδιση και ρύθμιση της ε, μετανάστευσης με αυτών των μεγαλών ροών των προσφύγων ε, έχουν να κάνουν με αντανακλαστικές κινήσεις, αλλά θα πρέπει πάνω απ' όλα να αφήσουμε αυτές τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν την ευρύτερη εικόνα. Αυτό ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το προσφέρει. Ξέρουμε ότι συζητούν τα κρατημένη προς την κατεύθυνση αυτή και κάτι ακόμη. Η δημιουργία νόμιμων ε, διόδων που ανέφερε η κυρία Κέντζ. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει νόμιμη δίωδος κατάρτισης για όλους, όχι μόνο τους πρόσφυγες, κατάρτισης, εκπαίδευσης. Αυτό δηλαδή πρέπει να ισχύει και για τους μετανάστες εργαζόμενους που ενδεχομένω εργάζονται παράνομα. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο θα λάβει ο εισηγητής κύριος Μπενιφέη. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος γιατί άλλωστε θα έχω αργότερα και τη δυνατότητα στην Επιτροπή μας να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Ωστόσο, ήδη από τώρα θα ήθελα να περάσω σε κάποιες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και να ευχαριστήσω όλους τους πυρογνώμονες και συναδέλφους που πήραν το λόγο. Νομίζω ότι η έκθεση πρωτοβουλίας μας θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο να θέσει το ζήτημα της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας ως πρόκληση και ως ευκαιρία κάνοντας μια συγκεκριμένη ανάλυση της κατάστασης, διευκρινίζοντας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα και κάνοντας συγκεκριμένε προτάσεις που να βασίζονται στις βέλτιστες υφιστάμενες πρακτικές. Θα πρέπει δηλαδή η πρόταση αυτή να ενθαρρύνει τη συζήτηση αλλά και την αντιπαράθεση με την κοινή γνώμη. Θα πρέπει και η κοινή γνώμη να εμπλακεί περισσότερο στο σημαντικότατο αυτό ζήτημα και στην όλη συζήτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχνάμε την οριζόντια προσέγγιση την οποία την τόνισαν πολλοί συνάδελφοι. Όντω αυτή τη στιγμή μέσω του προσφυγικού ζητήματο στίγονται πολλές επιμέρους πολιτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πάρα πολλά μέτωπα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ολιστική προσέγγιση της μετανάστευση στη Μεσόγειο, τη Εσίλ Κέγκε, γιατί το ζήτημα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής, το ζήτημα της μεταρρύθμισης των ε, υφιστάμενων κανόνων όπως τη σύμβαση του Δουβλίνου είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την επιτυχία της ένταξης των ε, προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το ζήτημα λοιπόν αυτό έχει να κάνει προφανώς με την απασχόληση αλλά παράλληλα θα πρέπει να προτείνουμε μεταρρυθμίσεις διότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες ακόμα και σήμερα δεν εφαρμόζουν την περίφημη οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής των μεταναστών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή και για ακριβώς αυτό το λόγο έχουμε μία κατάσταση που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλες αποκλήσεις και διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταυτού πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε μία κοινή πολιτική, κοινού όρους και συνθήκες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην χρησιμοποιούμε χρηματοδοτικούς πόρους που ήδη χρησιμοποιούνται για άλλες ευάλωτες ομάδες ή μη προνομίχες ομάδες. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε συνθήκες ανταγωνισμού ή συναγωνισμού τους Ευρωπαίους πολίτες και τους μεταναστές, τους πρόσφυγες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το μόνο που καταφέρνουμε κατά αυτόν τον τρόπο είναι να ενισχύσουμε τη ρατσιστική ρητορική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα θα πρέπει να αναλάβουμε θετική δράση για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Όπως το είπανε και πολλοί εμπειρογνώμονες, οι αγορές εργασίας στα κράτη-μέλη διαφέρουν. Επομένως χρειάζονται και διαφορετικές προσεγγίσεις που να λαμβάνουν υπόψη τους ακόμα και τις υφιστάμενες δεξιότητες επαγγελματικές που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή μια κοινή μαγική λύση για όλες τις χώρες η μεταρρύθμιση του συστήματος της μπλε κάρτας που η κυρία Κέγκ επίση ανέφερε είναι πολύ σημαντικό. Περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω όμως ότι και εμείς θα πρέπει να συμβάλλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, πρέπει να αναλάβουμε δράση προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις αιτήσει ασύλου. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να επιταχύνεται η όλη διαδικασία τη στιγμή που πάρα πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να ενταχθούν τελικά σε ένα γενικότερο καθεστώς διεθνούς προστασίας. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία αυτή, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να οδηγηθούμε σε μια αποτελεσματική ομαλή ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το ζήτημα της οικογενειακής ε, επανένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνδέεται με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και βέβαια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ληφθούν οι σωστές πολιτικές αποφάσεις. Τέλος, οι πόροι. Υπάρχουν διάφοροι, διάφορα ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Σύνταξης, έχουμε το Ταμείο για τα λιγότερα προνομιούχα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα διαφορετικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρα από τον καλύτερο συντονισμό και τις καλύτερες συνέργειες θα πρέπει και σε εθνικό επίπεδο να έχουμε επιχειρησιακά προγράμματα. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται με πολύ βραδείς ρυθμούς στα κράτη-μέλη και αυτό οδηγεί σε πολλές δυσκολίες. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε καλύτερες λύσεις και μάλιστα ευρωπαϊκές λύσεις. Και κάτι ακόμα, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο τους εμπειρογνώμονες και ακόμα περισσότερο τους συναδέλφους για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια θετική έκθεση το Μάρτιο. Προσβλέπω λοιπόν σε μια θετική ανταλλαγή απόψεων στον διάμεσο αυτό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρουσιάσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας και όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε. Δεν σταματάει εδώ αυτή η προσπάθεια, συνεχίζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ως ε, Επιτροπή Απασχόληση είναι να δημιουργούνται δουλειέ, να δημιουργούνται θέσει εργασία για να μπορεί ο κόσμο να εντάσσεται, να ενσωματώνεται στην κοινωνία και να αρχίζει μια νέα ζωή σε ένα άλλο μέρο του κόσμου. Θα επανέλθουμε και είμαι βέβαια ότι και άλλε επιτροπές θα εργαστούν επί των ιδίων θεμάτων. είναι ευρεία η πλειοψηφία, παρόλο που ακούγονται διάφορα σχόλια από διάφορες πλευρές και στη δική μας επιτροπή, πάντως υπάρχει ευρεία ε, πλειοψηφία που στο Κοινοβούλιο είναι πρόθυμη να αγωνιστεί έτσι ώστε αυτή η νέα Ευρώπη να λειτουργήσει σωστά. Που είναι άνθρωποι, που είναι άνθρωποι από άλλα μέρη του κόσμου και έρχονται κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε στη συζήτηση αυτή και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και βεβαίως πάντα μας ενδιαφέρει να έχουμε μόνιμη και διαρκή επαφή μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.